Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Έχουμε ήδη αρχίσει, αργήσει λίγο, γι' αυτό ζητώ πρώτα απ' όλα συγγνώμη εκ μέρους του Πρόεδρου, ο οποίος ε, λόγω απρόπτων δεν μπορεί να είναι εδώ. Σας καλωσορίζω μετά τις διακοπές και αρχίζουμε με μια από τις πιο σημαντικές μέρες για τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, γιατί πολλά από αυτά που θα συμβούν σήμερα δεν θα ξανασυμβούν για χρόνια ακόμα. Οπότε αρχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης πρώτα απ' όλα. Δεν βλέπω σχόλια. Ε, του Πρόεδρου δεν έχω. Θέλω όμως να σας ενημερώσω για το ότι το χρονοδιάγραμμα για τις συνεδριάσεις μας το 2020 που ενέκριναν τον Ιούλιο οι συντονιστές συμπεριλαμβάνεται στους φακέλους σας, οπότε κοιτάξτε το και αν δεν έχετε σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως θεωρείται εγκεκριμένο. Και πάμε στο σημείο 4. Και καλωσορίζω εδώ τον κύριο Ανδρέα Ενρία, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ποπτικού Συμβουλίου που δημιουργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα πλαίσια του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Ο κύριος Ενδρία ξεκίνησε την πεντετή του θητεία ως πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου την 1η Ιανουαρίου του 2019. Είναι η δεύτερη δημόσια ακρόαση που έχουμε μαζί του υπό την ιδιότητά του αυτή. Σήμερα θα συζητήσουμε μαζί σας μεταξύ άλλων και τα εξή. Τις προκλήσεις, τις ρυθμιστικές και τις εποπτικές που αντιμετωπίζετε, την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά την προετοιμασία για το Brexit και τι γίνεται ε, με την ε, Τραπεζική Ένωση και την καταπολέμηση της νομοποίησης ε, εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας και θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαδιοδότηση την εναρμόνιση κανόνων κλπ. Θα σας δώσουμε 10 λεπτά για την αρχική σας παρουσίαση και στη συνέχεια θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Για 5 λεπτά, όσο πιο σύντομη είναι η ερώτησή σας, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχει ο κύριος Ενρία για να σας απαντήσει. Ε, αν υπάρξει χρόνος θα πάμε και στο Catch αλλά στις 10.30 θα πρέπει να τελειώσουμε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε και άλλη σημαντική ακρόαση μετά. Χωρί άλλη καθυστέρηση λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Νερία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι και κύριοι βουλευτέ, είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ για αυτή την πρώτη ακρόαση ενώπιον του νέου εκλεγέντο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αποτελεσματικότητα του εποπτικού μα έργου και η συνέπεια των αποτελεσμάτων μα στην εποπτεία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο εναρμόνιση του ρυθμιστικού πλαισίου και τα σχόλια και η ανάδραση από ε, τον επόπτη για την καθημερινή εφαρμογή αυτών των κανόνων είναι θεμελιώδου σημασία για να το διασφαλίζει ότι οι στόχοι που τίθενται στην νομοθεσία τηρούνται ε, σε ένα ε, περιβάλλον αγοράς που συνεχώς αλλάζει. Η επιτυχία λοιπόν της Τραπεζικής Ένωσης εξαρτάται από την επικοδομητική μας συνεργασία. Η εποπτεία των τραπεζών της ΕΚΤ ε, έχει αναλάβει τη δέσμευση να πληρεί τα καθήκοντα λογοδοσία έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανεξαρτησία και λογοδοσία είναι θεμελιώδη για την υψηλή ποιότητα της εποπτείας και έχουμε βεβαίω δεσμευτεί να έχουμε καλή συνεργασία και με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατα συμφωνήσαμε με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ένα μνημόνιο συνεργασία για την πρακτική μα συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και θα υπογραφεί αυτό το μνημόνιο τον Οκτώβριο. Το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει αυτό το μνημόνιο συνεργασία, το οποίο θα διασφαλίσει ότι το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί να εκτελεί το ελεγκτικό του έργο για την εποπτεία τραπεζών τη ΕΚΤ. Δείχνει την καλή θέληση μεταξύ των δύο για την επικοδομητική μα συνεργασία του χρόνου, όπως και κάθε χρόνο, θα συνεχίσουμε να οργανώνουμε το έργο μας γύρω από κάποιες βασικές προτεραιότητες εποπτείας. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ε, μετά την κρίση θα συνεχιστεί, είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων, των προτεραιοτήτων μας και επίσης θα ασχοληθούμε με τους αναδυόμενους κινδύνους ε, για τα αίτια της χαμηλής ε, κερδοφορίας και της χαμηλής αποτίμησης αγοράς για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Ιδιαίτερος, θα συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με την καθοδήγηση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και με τις συστάσεις που προκύπτουν από την αναθεώρηση των εσωτερικών υποδειγμάτων και θα κάνουμε επιτόπου αποστολές για να ασχολούμεθα με τους εμπορικούς κινδύνους και τις αποτιμήσεις ενεργητικού. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε ε, τα κριτήρια ανάληψης ε, και πλήρους κάλυψης πιστώσεων ε, των τραπεζών και την ποιότητα των εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίων και ρευστότητα. Θα παρακολουθούμε την βιωσιμότητα των ε, επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών και ε, την κερδοφορία και την ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και θα παρακολουθούμε και το κατά πόσο είναι ευάλωτε οι τράπεζε σε θέματα τεχνολογία πληροφοριών και ε, κινδύνου ε, κυβερνοχώρου. Άλλα βασικά θέματα θα είναι τα stress και οι συνολικές αξιολογήσεις θα συνεχίζουν, ε, θα συνεχίζουν στους επόμενους μήνες λαμβάνοντα υπόψη και την μετατόπιση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των τραπεζών στην Ευρωζώνη ω συνέπεια του Brexit και καθώ ε, τα κράτη-μέλη όπω η Βουλγαρία και μετά η Κροατία ζητούν στενότερη συνεργασία. Τώρα θα ήθελα να μιλήσω για κάποια από τα βασικά θέματα που ε, μα έχουν απασχολήσει του τελευταίου μήνε. Όπω θα θυμάστε, η Εποπτεία Τραπεζών τη ΕΚΤ ε, είχε αναλάβει να επαναξετάσει τι απαιτήσει για την εποπτεία όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Τώρα έχουμε αξιολογήσει την σχέση μεταξύ της δικής μας προσέγγισης ε, και ε, του νέου πυλώνα ένα για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, όπως ε, παρατίθεται στον τελευταίο κανονισμό για τις κεφαλιακές απαιτήσει και έχουμε καταλήξει ότι χρειάζονται κάποιες προσαρμογές στις απαιτήσει μας, ε, στις προβλέψεις προληπτικής εποπτείας ε, για τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Αυτές οι προσαρμογές θα ενισχύσουν την συνέπεια και απλούστευση της συνολικής μας προσέγγισης και θα μειώσουν τον βάρος υποβολής εκθέσεων ε, από πλευράς τραπεζών. Οι απαιτήσει ε, εποπτείας της ΕΚΤ για τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα περιορίζονται σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα τα οποία προκύπτουν από δάνεια πριν τι 26 Απριλίου του 2019 που δεν υπόκεινται ε, σχέδιο ε, του πυλώνα 1. Ε, Μετά τι 26 Απριλίου 2019, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα υπόκειται σε αυτές ε, τις νέες διατάξεις. Οι απαιτήσει εποπτεία για τα παλαιότερα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, δηλαδή αυτά τα οποία είχαν ταξινομηθεί ω μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στι 31 Μαρτίου του 2018, δεν έχουν τροποποιηθεί, όπω έχουν ανακοινωθεί στι επιστολέ SREP που εστάλησαν στι τράπεζε και σε ένα ανακοινωθέν που δημοσίευσε η ΕΚ τον Ιούλιο του 2018. Από την προηγούμενη ε, ακρόασή μου ενώπιν τη Επιτροπή σα, έχουμε συνεχίσει να προετοιμάζουμε την ετοιμότητα των τραπεζών για τον Brexit, καθώ και την πιθανότητα ενός σενάριου μη συμφωνίας το οποίο συνεχίζει να μας ανησυχεί. Έχουν ληφθεί μέτρα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις ε, για να είναι προετοιμασμένος ο ιδιωτικός τομέας για το ενδεχόμενο της μη συμφωνίας. Οι τράπεζες θα επιταχύνουν την υλοποίηση των σχεδίων τους για τον Brexit, για, να είναι πλήρως προετοιμασμένες στην περίπτωση ενός Brexit χωρίς ε, συμφωνία στο τέλος Οκτωβρίου. Τώρα, ας μιλήσω για κάποιες ρυθμιστικές προκλήσεις για τον τραπεζικό τομέα, για την καινούργια θητεία. Στην παρούσα συγκυρία είναι σημαντικό να θυμηθούμε τα διδάγματα από την τελευταία κρίση. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την πλήρη εφαρμογή τη Βασιλεία 3. Ο κύκλο μεταρρυθμίσεων πρέπει να ολοκληρωθεί και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το σημαντικό έργο που έχουμε ξεκινήσει. Πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο μα για τα ενεργητικά σταθμισμένα ω προ τον κίνδυνο και για τα εσωτερικά υποδείγματα. Ο στόχο είναι να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζε οι οποίε στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν τα εσωτερικά υποδείγματα για να μειώσουν ε, το ρυθμιστικό του κεφάλαιο, θα πρέπει να κάνουν τι απαραίτητε ε, προσαρμογές. Τα διεθνή ε, πρότυπα ε, αντικατοπτρίζουν τις αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και τη συνέπεια των σταθεσμένων ενεργητικών ε, σύμφωνα με την αναθεώρηση των εσωτερικών υποδειγμάτων ε, της ΕΚΤ. Επίσης, θα πρέπει ε, να αναγνωρίσουμε ότι η υλοποίηση του αποτελέσματος τυποποιημένων προσεγγίσεων της Βασιλείας 2 ήταν επίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα το νέο αποτέλεσμα είναι πιο δαπανηρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι σε άλλες δικαιοδοσίες. Και παρότι το αποτέλεσμα των τυποποιημένων προσεγγίσεων μπορεί να έχει ένα δικαιολόγητο αντίκτυπο σε επιχειρηματικέ δραστηριότητε χαμηλού κινδύνου, διασφαλίζει πιο δίκαιο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών που χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα και τραπεζών που βασίζονται σε τυποποιημένη προσέγγιση. Είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε το τελευταίο κεφάλαιο τη μεταρρύθμιση μετά την κρίση. Μετά την υλοποίηση τη Βασιλεία 3, η επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού και τη οδηγία ε, κεφαλαιακών απαιτήσεων πρέπει να αποτελέσουν μια ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε τι τις, απαιτούμενες, τις υπάρχουσες ε, ελλείψεις. Ε, επιπροσθέτως, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν από τα ε, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να πληρούν τις απαιτήσει του πυλώνα 2 με ε, κεφαλαιακά εργαλεία υψηλής ποιότητας, το κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1. Όσον αφορά τις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την θεσμική αρχιτεκτονική της Τραπεζικής Ένωσης, όπου λείπει ο τρίτος πυλώνας, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Τα διαφορετικά εμπόδια για την ολοκλήρωση και ενοποίηση τραπεζών που προκαλούνται από την μη ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης μαζί με άλλα νομοθετικά εμπόδια για τις ε, διασυνοριακές δραστηριότητες τραπεζών στην Ευρωζώνη ε, επηρεάζουν ε, την υγιή δραστηριότητα των τραπεζών μας που πλήττονται από τις χαμηλές αποτιμήσεις της αγοράς. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι στο, στην προληπτική μας εποπτεία ενσωματώνουμε και την, το θέμα της αντιμετώπισης της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Ε, η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και με τις εθνικές, εθνικές εποπτικές και προληπτικές αρχές ε, που ασχολούνται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος και χρήματος ε, από τρομοκρατικές δραστηριότητες και η λειτουργία συντονισμού ε, του ε, SSM καθοδηγεί το εσωτερικό έργο που γίνεται και προσαρμόζει τη μεθοδολογία του SSS ώστε να λαμβάνει υπόψη ε, τα θέματα που έχουν σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία συχνά συζητούσαμε και με τον προκάτοχό μου και με την Επιτροπή αυτή κατά τους τελευταίους μήνες, κατά την τελευταία θητεία. Μεταξύ αυτών ε, είναι ο δανεισμός υψηλού κινδύνου, τα stress tests και τα εσωτερικά υποδείγματα. Εμείς παρέχουμε προληπτική ε, καθοδήγηση και εποπτική καθοδήγηση για το δανεισμό υψηλού κινδύνου, αλλά πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση για τις εξελίξεις της αγοράς, γιατί η αγορά ε, αλλάζει ταχύτατα και θα συνεχίσουμε όπως έχουμε ήδη διεξαγάγει στοχευμένα stress test για να ε, επανεξετάσουμε τον κίνδυνο ρευστότητας και προετοιμάζουμε ήδη stress test για τον επόμενο χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα εσωτερικά υποδείγματα το έργο μας ήταν αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση ε, κάποιων ελλείψεων και των αδικαιολόγητων διαφορών στο πώς χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα οι τράπεζες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ενρία και θέλω να Καταλάβω ότι έχουμε ε, ε, λίγο χρόνο για τις ερωτήσεις. Παρακαλώ να είναι σύντομες οι ερωτήσεις για να μπορούν να δίνονται απαντήσεις. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είναι μεγάλη χαρά για μας που είστε κοντά μας ε, και θα κάνω σύντομες ερωτήσεις. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά τη Συμφωνία Βασιλεία 3, γιατί το αναφέρατε. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αποκλίνει και γιατί από τη συμφωνία αυτή. Το δεύτερο ερώτημά μου αφορά τα ΣΡΕΠ τη διαδικασία επιπτικού ελέγχου και αξιολόγηση. Εσείς έχετε αντιμετωπίσει κάποιο είδος κινδύνου ε, σε συγκεκριμένους τομείς όπου ισχύουν αυτές οι διαδικασίες ΣΡΕΠ. E ε, όσον αφορά το Brexit, ξέρετε ότι ο μηχανισμός σταθεροποίησης πιέζει τις τράπεζες ε, να εφαρμόζουν έκτακτα μέτρα. Ε, όλα αυτά τα γνωρίζουμε, αλλά πρόσφατα επισημάνατε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει περαιτέρω προσαρμογή των λογιστικών, των τραπεζών. Δεν υπάρχει όμως αρκετός χρόνος για να το επιτύχουμε αυτό. Ε, βλέπετε λοιπόν υπάρχουν δυνατότητες έτσι ώστε να επιτευχθεί ε, κάποια επιτυχία στους επόμενους 1,5, ε, στον επόμενο 1,5 μήνα. Και κάτι άλλο, κυρία Νουή, θέτει το θέμα των εθνικών επιλογών, των ε, αποφάσεων. Ορισμένες από αυτές έχουν εντοπιστεί και ένα από τα θέματα είναι τα εθνικά καθεστώτα πτώχευσης. Εσείς ε, πιστεύετε ότι οι νομοθέτες Ευρωπαϊκή Ένωσης θα μπορούσαν να προσφέρουν κάτι σε αυτή την κατεύθυνση και βλέπετε να υπάρχει κάποια δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ε, η εμπειρία και, το πολύ, και η πολύ πλούσια εργαλειοθήκη που έχουν οι Αμερικανοί για τέτοιου περιπτώσει τη δυνατότητα να μάθουμε από τους Αμερικανούς αυτό το θέμα. Πάρα πολύ ωραίες, πολύ πλούσιες ερωτήσεις για να απαντήσω. Θα έπρεπε να έχουμε μια ολόκληρη μέρα. Θα προσπαθήσω να είμαι ε, πιο σαφής, αλλά θα προσπαθήσω να μπω και σε λεπτομέρειες ε, της ερώτησης. Όσον αφορά τη Βασιλεία 3 για απόκληση από τις διεθνείς προδιαγραφές, να σας πω ότι οι περισσότερες προτάσεις που έχουν κατατεθεί και αφορούν στα διεθνή πρότυπα είναι σε απόλυτη συμφωνία με την ανάλυση που έχει γίνει από την ΕΚΤ, με τις ε, προτάσεις της ΕΚΤ και με τα πορίσματα των δικών μας των αναλύσεων των εσωτερικών προτύπων, ε, των εσωτερικών υποδειγμάτων. Άρα δηλαδή ε, πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία αναθεώρησης που για μένα είναι πολύ σημαντική. Δεν βλέπω να υπάρχει κανένας λόγος για απόκληση και επιπλέον αν δείτε τις επιπτώσεις θα δείτε ότι η προσαρμογή είναι κυρίως στις μεγάλες τράπεζες. Αν θυμάμαι καλά, οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την είναι περίπου 135 δις και 127 εξ αυτών ε, είναι ε, συστημικέ ε, τράπεζε, πολύ σημαντικέ σε παγκόσμιο επίπεδο και άλλα συστημικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Άρα δηλαδή μιλάμε για μεγάλε διεθνεί τράπεζε. Ω εκ τούτου η ιδέα των να υπάρχουν ιδιαιτερότητε για αυτέ τι ε, τράπεζε, κατά την άποψή μου δεν είναι επιθυμητό. Το μόνο θέμα το οποίο με απασχολεί σχετικά με το πακέτο τη Βασιλεία είναι το επίπεδο εκρών, output floor. Αυτό είναι ένα αίτημα που έχει κατατεθεί από πάρα πάρα πολλές ε, ε, νομολογίες και τράπεζες και ιδρύματα που δεν εξαρτώνται από τα εσωτερικά υποδείγματα. Έχουμε κάνει κάποιες διαδικασίες ε, μέσα από αυτή τη διαδικασία της ΕΚΤ βλέπω να υπάρχει το ενδεχόμενο στρεβλώσεων που θα μπορούσε να προκαλέσει και κάποια ευαισθησία. Παράλληλα όμως αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τουλάχιστον όσον αφορά ε, στα διεθνή πρότυπα. Πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας ε, στην διεθνή κοινότητα. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα που δείχνουν ότι θα πρέπει να είμαστε πιστοί στις διαπραγματεύσεις μας θεωρώ ότι δεν θα πρέπει όλα αυτά να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για τις τρέπεζες. Για το δεύτερο ερώτημά σας, πράγματι υπάρχουν θέματα συγκέντρωσης ε, κινδύνων. Αλλά το βασικό θέμα που θέλω να σε επισημάνω είναι ότι υπάρχουν ενδεχομένως μόνο δύο τομείς όπου, τα, όπου οι ΣΡΕΠ θα μπορούσαν να προκαλέσουν ε, κάποια επιδείνωση, ε, η κίνδυνη διαχείρισης και λειτουργίας. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Τα θέματα της διαχείρισης, της διακυβέρνησης έχουν προκύψει, υπάρχουν θέματα AML για το ξέπλυμα χρήματος. Όσον αφορά το λειτουργικό, πρέπει να σας πω ότι σε πάρα πολλές έρευνες που έχουμε κάνει, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν απάτες που έχουν σχέση με τις υποδομές, με τα δεδομένα, αλλά και με την πρόκληση της ε, ψηφιοποίησης, αλλά και στον, στην κυβερνοαπειλή και εκεί πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Όσον αφορά το Brexit, πράγματι ε, στα μηνύματά μας ε, από ευρωπαϊκής πλευράς έχουμε επισημάνει ότι πρέπει να ε, είναι πιο ουσιαστικά τα business models. Ε, αυτό το είπαμε σε όλους όσους μας πλησίασαν για ερωτήματα κατάσταση. Και είπαμε ότι όσον αφορά τα στοχευμένα μοντέλα που έχουν ορίσει οι τράπεζες ε, και που έχουν συμφωνηθεί με μας, εκεί πράγματι φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνη διαχείριση στην Ευρωζώνη. Αυτό που είπα στι αρχικέ μου παρατηρήσει. το βασικότερο είναι το θέμα τη εκτέλεση. Βλέπουμε ότι ενώ έχει συμφωνηθεί το θέμα του δανεισμού, το πόσο γρήγορα προχωράει κανεί ε, προ τα εκεί και τα βήματα που πρέπει να γίνουν, ε, επ' αυτού είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί, γιατί δεν υπάρχει ικανοποιητική πρόοδος. Όσον αφορά την εθνική διακριτική ευχέρεια, ε, κυρίως για θέματα πτωχεύσεων, Κοιτάξτε για τις πτωχεύσεις, έχουμε εκεί ένα πρόβλημα. Αυτό που υπάρχει είναι ότι στο BRD υπάρχει η παραδοχή ε, ότι η ΕΚΤ είναι εκείνη που ορίζει μια τράπεζα αν θα πτωχεύσει ή όχι και κατόπιν αν το θέμα ε, περνάει σε μια εθνική διαδικασία ε, καθάρισης. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι απαραίτητο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ασχοληθούμε με το τι θα συμβεί αργότερα. Η εμπειρία όμως που έχουμε κάνει είναι ανησυχητική. Έχουμε τράπεζες ε, οι οποίες ε, ε, θα έπρεπε να πτωχεύσουν, αλλά δεν μπαίνουν σε καθάριση, γιατί δεν υπάρχει ε, νομική βάση. Όπως στη Λετωνία, εκεί είδαμε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ως εκ τούτου αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα παραμένει με την άδειά της για μεγάλο χρονικό διάστημα, άσχετα αν είναι σε κινδυνεύουμε πτώχευση ή όχι και μόνο σε περιπτώσεις όπου έχουμε κανονικές διαδικασίες ε, πτώχευσης, μόνο εκεί μπορεί να υπάρξει εξέλιξη, δηλαδή να υπάρξει και κρατική ε, αρρωγή. Νομίζω λοιπόν ότι το θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση σε αυτό το τομέα και εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχουν διοικητικά εργαλεία για την πτώχευση, κάπως όπως τα έχουν ρυθμίσει οι Αμερικανοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον χρόνο, ε, να υποβάλλετε και ερωτήσεις που θα μπορούν να σας απαντήσουν μέσα ε, σε πέντε λεπτά. Ε, Φερνάντες για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ισπανικά. Πρώτα απ' όλα, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας αυτή. Και θέλω να σας ρωτήσω μετά από την κυρία Χούμπνερ, που ουσιαστικά υπέβαλε πολλές από τις ερωτήσεις που θέλαμε και εμείς να υποβάλουμε. Δύο πράγματα λοιπόν εγώ θέλω να ρωτήσω. Το ένα είναι την διαδικασία εισόδου της Βουλγαρίας και της Κροατίας στην Τραπεζική Ένωση. Έγκριση του ευρώ και διεύρυνση ώστε να συμπεριληφθεί και στον εποπτικό μηχανισμό. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω εσείς τη διαδικασία αυτήν πώς τη βλέπετε. Πώς βλέπετε το χρονοδιάγραμμα. Πότε μπορούμε να ελπίσουμε ότι δύο αυτές χώρες θα ενταχθούν στο ευρώ. Και σε τι βαθμό η διαδικασία αυτή μπορεί να αποτελέσει και παράδειγμα για άλλες χώρες οι οποίες βρίσκονται εκτός ευρώ σήμερα και που όπως λένε και οι συνθήκες κάποια στιγμή μπορούν να ενταχθούν. Δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τα προβλήματα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Στην Επιτροπή μας σε λίγο έχουμε ακρόαση με την υποψήφια για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Επιτροπής. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι η κατάσταση της νομισματικής ε, πολιτικής ε, προσφοράς χρήματος να συνεχιστεί σύμφωνα βέβαια με τις προοπτικές που βλέπουμε στην Ευρωζώνη και ανάλογα με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε και τους επόμενους μήνες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τι επιπτώσεις θα έχει στην σταθερότητα αν υπάρξει περισσότερο επεκτατική πολιτική από πλευρά σας στην ε, δημοσιονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας για το θέμα της στενής συνεργασίας. Το αίτημα δηλαδή από τη Βουλγαρία και την Κροατία για στενή συνεργασία μαζί μας. Πράγματι βρισκόμαστε στην διαδικασία ολοκλήρωσης της ε, συνολικής αξιολόγησης για τις βουλγαρικές τράπεζες και έχουμε τοπίσει δύο τράπεζες που δεν έχουν ε, αρκετή κεφαλοποίηση και θα έπρεπε να διορθωθεί αυτό. Τώρα λοιπόν είμαστε στην διαδικασία παρακολούθησης ε, των τραπεζών αυτών που σχεδιάζουν για να καλύψουν τα, τις διαφορές, τα ελλείμματα και να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τα σχέδια αυτά, οπότε εφόσον γίνει αυτό θα αναλάβουμε και τα επόμενα βήματα στη διαδικασία που είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας ουσιαστικά και μετά να μπούμε σε αυτήν την στενή συνεργασία. Και αυτό έχει να κάνει και γενικότερα με την ένταξη στο ευρώ που θα αρχίσει τότε. Με την ε, Κροατία θα ξεκινήσουμε την αξιολόγηση πολύ σύντομα, τώρα το Σεπτέμβριο νομίζω. Γενικά είδαμε στη βουλγαρική περίπτωση ότι ένας χρόνος περνάει από τη στιγμή που υποβάλλεται το αίτημα και ολοκληρώνεται η αξιολόγηση με αίτημα για κεφαλοποίηση εφόσον υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Λίγο πολύ δηλαδή το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι. Βέβαια η διαδικασία εξαρτάται και από την ε, ε, νομική κατάσταση, από τις λεπτομέρειες. Και αυτό έγινε στην περίπτωση της Βουλγαρίας και θα γίνει με την Κροατία για να είμαστε σίγουροι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα ύδατα. Αυτή δηλαδή η συνεργασία είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας. Όσον αφορά την νομισματική πολιτική, ξέρετε ότι υπάρχει η διάκριση. Νομισματική πολιτική από τη μια μεριά, υποπτή από την άλλη. Όμως, στο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που έχουμε τώρα για αρκετό καιρό, πιέζει προς τα κάτω τα διατραπεζικά περιθώρια και από την άλλη μεριά μακροοικονομικά υπήρξαν βελτιωμένες προπτικές που βελτίωσαν και τη δυνατότητα των δανειστών να πληρώσουν τα δάνειά τους και άρα και τις τράπεζες να έχουν λιγότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και υπάρχει και θετική επίπτωση στους όγκους. Πώς θα τα ισορροπήσουμε αυτά, αυτό είναι ένα ζήτημα. Επιτρέψτε μου να πω επίσης ότι υπάρχει και το θέμα της μακροπροληπτικής πολιτικής. Οπότε όταν έχουμε προσφορά χρήματος αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποιους ε, κινδύνους. Οι επενδυτές, οι τράπεζες μερικές φορές αρχίζει η ενίσχυση της μακροπροληπτικής προστασίας τότε. Ευχαριστούμε. Λουί Καριγκάνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ενερία που ήρθατε εδώ. Υπάρχει πάντα ο φόβος της ύφεση που αυξάνει στις αγορές τελευταία. Οπότε η ερώτησή μου είναι τι γίνεται με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επ' αυτού δύο ερωτήματα. Πρώτον, για το Doom Loop, τη δυνατότητα να επιστρέψει. Η έκθεση τα κρατικά ομόλογα. Ο κίνδυνος εδώ είναι ιδιαίτερα υψηλός. Υπήρξε μία πρόταση ότι η έκθεση της Επιτροπής έχει να κάνει με τα security κυρίως και η Επιτροπή έκανε μία πρόταση, εμείς είμαστε στη δικασία πρώτης ανάγνωσης και δεν βλέπουμε να προχωράει στο Σεβούλιο καθόλου το θέμα. Λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, πόσο σημαντικό είναι να υιοθετηθεί η πρόταση αυτή. Βλέπετε μήπως και άλλα μέσα να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πόσο θα μπορούσε να συνεισφέρει το Εποπτικό Συμβούλιο. Δεύτερον, για τη μείωση κινδύνου, που είναι και αυτό ένα πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Εσείς Πιστεύετε ότι πρέπει να περιμένουμε ώστε να υπάρξει μείωση κινδύνου πριν υιοθετήσουμε μέτρα επιμερισμού κινδύνου. Τι πρόοδος έχει γίνει επίσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ποια είναι η άποψή σας για το κατά πόσον τώρα θα ήταν δυνατόν, εσείς θα το συμβουλεύατε, υπάρχουν οι προϋποθέσεις να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε ένα backstop για τον ενίο μηχανισμό εξυγένσης. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Όσον αφορά τους φόβους για ύφεση. Όντως, σκοτεινιάζει ο ουρανός και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Θέλω όμως μόνο να υπενθυμίσω ότι πρόσφατα κάναμε τις δοκιμές αντοχής που είδαμε ότι έχει ενισχυθεί η αντοχή. Υπήρξαν τέτοια αποτελέσματα που δείχνουν ότι υπάρχει αντοχή. Όμως υπάρχει χαμηλή κερδοφορία, υπάρχει χαμηλή ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου, πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Το Ντούμλουπ τώρα και το θέμα της έκθεσης η ευρωπαϊκή εποπτεία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Αλλά δεν μπορούμε από μόνοι μας να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο εντοπίστηκε στην ε, πρόσφατη κρίση. Το είδαμε αυτό με τα κρατικά ομόλογα και κατά πόσο οι τράπεζες ήταν σε θέση με λογικές συνθήκες να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα. Επιτρέψτε μου να πω λοιπόν πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν εποπτικά μέσα για να ελεγχθεί η έκθεση των τραπεζών σε κρατικά ομόλογα. Και στις δοκιμές ε, αντοχής το κοιτάζουμε αυτό και βλέπουμε τη δυνατότητα των τραπεζών να αντέξουν. Όταν δούμε ότι υπάρχει υπερβολική συγκέντρωση τέτοιας έκθεσης, τότε μπορούμε να αναλάβουμε δράση. Εγώ προσωπικά πάντα στήριζα πάρα πολύ την πρόταση SSBS, που είναι πρόταση που έρχεται και από την Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή του SRB και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο τα δύο πράγματα πάνε μαζί. Δηλαδή το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εκθέσεις αυτές να είναι καλύτερο και συγχρόνως να υπάρχει, πώς το πω, μια ε, κοινή λογική που να αναπτύσσεται. Έτσι αλλιώς τα μέσα που διαθέτουμε είναι γνωστά. Ένα από τα στοιχεία κλειδί εδώ είναι η σύνδεση με την αγορά. Βλέπουμε ότι οι τράπεζες όταν έχουν τέτοια μεγάλη έκθεση κρατικά ομόλογα αλλάζουν την στάση τους. Ε, φροντίζουν να υπάρχει κάποια πειθαρχία και νομίζω ότι αποτελεί και κίνητρο για τις τράπεζες να περιορίζουν την έκθεσή τους αυτή. Τώρα για την εκτίμηση κινδύνου και τον επιμερισμένο κίνδυνο. Ήδη από το 2018 Είμαστε κάτω από 50 δισεκατομμύρια ε, τιτλοποίησης ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οπότε υπάρχουν κατασχέσεις, υπάρχει τιτλοποίηση, πάντως τα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων πέφτουν. και οι τράπεζες ε, καταφέρνουν σιγά σιγά να πετύχουν το στόχο τους. Πετυχαίνουν το στόχο που έχουμε συμφωνήσει μαζί τους δηλαδή. Τώρα, το ότι πρώτα πρέπει να κάνουμε κάτι και μετά πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς πάντα λειτουργούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με χάρτες πορείας. Όταν πρέπει να υπάρχει διόρθωση, πρέπει να υπάρχει διόρθωση. Και έτσι σιγά σιγά προχωράμε. Ευχαριστούμε εκ μέρους των Πρασίνων, ο κύριος Γκίγκολτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το μήνυμα το, οποίο ακούω από εσά, Ανδρέα, και από την έκτη γενικότερα είναι το εξής. Αφενός μεν, το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρώπη επιδεινώνεται, αλλά οι τράπεζες είναι καλύτερα προετοιμασμένες. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε την ΕΚΤ από την νομισματική πλευρά να κοινώνει χαμηλά επιτόκια και θα συνεχίσει να είναι κάπως ε, ακτιβιστική από πλευράς νομισματικής πολιτικής. Αυτό και για τις τράπεζες και για άλλους ε, φορείς της αγοράς με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Θεωρείτε ότι θα πρέπει οι εποπτικές αρχές να αυξήσουν τις προσπάθειες ώστε τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν να έχουν κοινέ δημοσιονομικές πολιτικές και να ενθαρρύνεται περισσότερο τις κοινέ οικονομικές πολιτικές για να μειωθούν οι πιέσει στα μακροπρόθεσμα ε, επιτόκια. Γιατί βλέπω πραγματικά κίνδυνο για τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. Δεν μπορεί ε, να στείνει προστατευτικά φράγματα μόνο έναντι μια τέτοια πορεία. και εδώ βλέπω και ένα ρόλο για την εποπτική πλευρά. Μπορεί η εποπτική πλευρά να καταστήσει σαφέ το τι πρέπει να κάνουμε για την κερδοφορία ε, και τον δανεισμό των τραπεζών. Θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα τη θέση σας επ' αυτού. Την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει, αλλά και στην εργασία σας στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, ε, ήσασταν υπέρ της διαφάνειας στην εποπτεία των τραπεζών. Μπορείτε να μας πείτε πόσο έχετε επιτύχει, θα ανακοινώσετε τα αποτελέσματα των stress test στην ΕΚΤ κάνετε και εσωτερικά stress test. Θα δημοσιεύσετε κατευθυντήριες γραμμές για τον πυλώνα 2 και θα μας δώσετε κάποια κλίμακα για αυτή τη γραφική παράσταση που έχετε κάνει με τις 107 τράπεζες, που όμως δεν έχει κλίμακα. Και επομένω, ε, δεν μπορούμε ούτε ανώνυμα να δούμε την κατανομή των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αυτή η γραφική παράσταση μπορεί να είναι η πρώτη γραφική παράσταση που θα δείξει τη διαφάνεια του κυρίου Ένρια, αν το βελτιώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώ από την τελευταία ερώτηση που νομίζω εύκολα μπορώ να σας απαντήσω θετικά. Μπορώ να δεσμευθώ υπέρ της μεγαλύτερης διαφάνειας και να κάνουμε και αυτή τη γραφική παράσταση πιο διαφανή. Επομένω, εδώ έχετε μια επιτυχημένη απάντηση. Τώρα, για τις απαιτήσει πυλώνα 2 και την αποκάλυψη αυτών των απαιτήσεων, δεν είμαι ικανοποιημένος με την φυστάμενη κατάσταση. 118 είναι οι τράπεζες, 76 ανακοινώνουν απαιτήσει πυλώνα 2, οι άλλες όχι. Έχουμε και διαφορετικές προσεγγισει όσον αφορά τι ρυθμιστικε απαιτήσει στην αγορά αξιογράφων. Προσπαθούμε και με την ΕΣΜΑ να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε πιο μεγάλη εναρμόνιση. Σίγουρα η νομοθεσία μας βοηθάει Ε, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, η νέα οδηγία CRD ε, θα απαιτεί από τις τράπεζες ε, να δημοσιοποιούν τις απαιτήσεις του πυλώνα 2 και αυτό θα είναι χρήσιμο. Για το B2G Έχουμε κάποιες εσωτερικές συζητήσεις, Υπάρχει κάποια, υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί ε, που έχουν ως αποτέλεσμα το ότι υπάρχουν αλλαγές στην προσέγγιση μας στον πυλώνα 2 γενικότερα, δηλαδή αναθεωρούμε την προσέγγιση στον πυλώνα 2, προσπαθώντας να το κάνουμε περισσότερο ανά συγκεκριμένο κίνδυνο και να χρησιμοποιούμε καλύτερα ό,τι στοιχεία έχουμε από τα iCaps και iLabs. Και ε, ο χρονικός προγραμματισμός αυτής της μετάβασης είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι μια ανησυχία, όχι δική μου προσωπικά, αλλά στην ε, εποπτική κοινότητα υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι αν αποκαλύψουμε τον το πυλώνα 2, οι αγορέ θα το θεωρήσουν ω σκληρέ ελάχιστε απαιτήσει που δεν είναι, γιατί αυτού του είδου τα προστατευτικά όρια υπάρχουν για να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε σε περίπτωση που τα χρειαστούμε. Το ερώτημά σα για την νομισματική πολιτική και πάλι ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η αρχή του ισχυρού διαχωρισμού, του αυστηρού διαχωρισμού και η θέση μου είναι ότι γενικά εμεί είμαστε ε, οι εποπτικέ αρχέ, αλλά και εμεί και οι τράπεζε Πρέπει να θεωρήσουμε την νομισματική πολιτική ως δεδομένη, ως εξωγενή παράγοντα και πιστεύω ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία για να λάβουμε υπόψη την πιθανή επίπτωση που θα έχει αυτό στην ανάληψη κινδύνων, στη στάση των τραπεζών για την ανάληψη κινδύνων ότι, ώστε τα μακροπροληπτικά προστατευτικά όρια θα πρέπει να υπάρχουν για να μην μπορέσουν κάποιες ακραίες νομισματικές πολιτικές να δημιουργήσουν υψηλούς κινδύνους. Και όσον αφορά την κερδοφορία πρέπει να πιέσουμε τις τράπεζες να αλλάξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα για να γίνουν πιο κερδοφόρες. Υπάρχουν αρνητικά επιτόκια σε άλλες χώρες. Στην Ελβετία, παραδείγματος χάρη, οι τράπεζες έχουν υψηλότερη κερδοφορία. Άρα υπάρχουν μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες για να βελτιωθούν. Τώρα, συγγνώμη που ξεπερνώ το χρόνο μου, αυτό που με ανησυχεί είναι ότι υπάρχουν διαρθρωτικά εμπόδια που δυσκολεύουν τις τράπεζες. Και αυτά τα διαρθρωτικά εμπόδια είναι η κατάτμιση της εσωτερικής μας αγοράς, της Τραπεζικής Ένωσης δηλαδή. Και αυτό εμποδίζει και την ενοποίηση και δεν επιτρέπει τις τράπεζες να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ πρέπει να ε, ε, εντοπίσουμε τις προσπάθειές μας. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα που θα το ε, εκφράσω με δύο τρόπους, λέει ο κύριος Ζουάν. Πιστεύετε ότι η διαδικασία εναρμόνισης και συγκέντρωσης θα καταλήξει ότι θα μείνουν μόνο κάποιοι συστημικοί όμιλοι στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αγορά. Και ε, θέτω την ερώτησή μου τώρα και με διαφορετικό τρόπο. Ε, η εναρμόνιση του συστήματος κινδύνων και η διαφορά μεταξύ των τραπεζών που είναι συνεταιριστικές, ε, που είναι περιφερειακές ή που είναι δημόσιες ε, θα, είναι, θα έχουν διαφορές. Εγώ θεωρούσα ότι η διαφοροποίηση των τραπεζών είναι παράγον αντοχής και θεωρούσα ότι το ότι δεν θα υπάρχουν πια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών τραπεζών και οι διαφορές μεταξύ καταστατικών των τραπεζών είναι, είναι παράγον αντοχής για το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Δηλαδή, η διαφοροποίηση στο οικοσύστημα του τραπεζικού τομέα είναι όντως ένα στοιχείο ισχύος και αντοχής. Και το έργο μας δεν το θεωρώ στοιχείο ε, τυποποίησης. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο για όλους και η αναλογικότητα είναι και μια ε, συνταγματική αρχή για την εποπτεία μας. Έχουμε καθορίσει την εποπτική μας προσέγγιση ανάλογα με την κλίμακα και ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο ε, των τραπεζών. Παρακολουθούμε με διαφορετικό τρόπο διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και εφαρμόζουμε απαιτήσει που αποτυπώνουν τι συγκεκριμένε ιδιαιτερότητε των τραπεζών. Εκεί όπου θέλουμε τυποποίηση είναι εκεί όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν βέλτιστε πρακτικέ και θέλουμε να ανεβάσουμε τον πύχη για όλε τι τράπεζε για να βελτιώσουμε την απόδοσή του. Να σα δώσω ένα παράδειγμα αν πάτε σε μια μικρή συνεταιριστική τράπεζα, μπορείτε να εφαρμόσετε αναλογικά απαιτήσει για την υποβολή εκθέσεων ή για την ανάγκη δημιουργίας συγκεκριμένων εσωτερικών επιτροπών κλπ. Αλλά τα επίπεδα διαχείρισης κινδύνου θέλετε να είναι στο σωστό επίπεδο. Θέλετε να υπάρχουν ε, έλεγχοι ε, για να υπάρχουν καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου. Σε πολλές δικαιοδοσίες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σκέφτονται να μην έχουν καθόλου την έννοια των σταθμισμένων ενεργητικών με βάση τον κίνδυνο. Εγώ δεν θα συμφωνούσα καθόλου με το να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοια προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι οι μικρές τράπεζες πολύ συχνά ε, δρούν κάπως ε, μαζικά για να αντιδράσουν σε συστημικούς κινδύνους. Επόμενος ε, για το ECR, ο Dirk Πέντινγκ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στο ότι ο ουρανός σκοτεινιάζει και νομίζω ότι καλό είναι να βλέπει κανείς και το μετρολογικό δελτίο τα θέματα που χειριζεστε είναι η Deutsche Bank, η οποία είναι καθαρά συστημική, είναι γιγαντιαία, αλλά με μια αδιευκρίνηστη δομή και γι' αυτό ερωτώ, σκέπτεστε να αναδιαρθρώσετε την Deutsche Bank. Ε, φαντάζομαι θα κατανοείτε ότι δεν μπορώ σήμερα εδώ να αναφερθώ σε μεμονωμένες τράπεζες. Φοβάμαι λοιπόν ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Λυπάμαι πάρα πολύ. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εάν υπάρχει κάτι που μπορώ να σας πω, είναι ότι θα πρέπει να ανησυχούμε για το ότι στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα μετά την κρίση δεν υπήρξε αρκετή και ικανοποιητική αναδιάρθρωση των τραπεζών. Γιατί αν συγκρίνετε τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα με αυτόν της Αμερικής, Νομίζω ότι η σύγκριση αυτή θα πρέπει να εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα των τραπεζών ε, είναι πολύ πιο ταχύς και γρήγορος. Ε, αντιμετωπίζονται πολύ πιο γρήγορα τα θέματα των κεφαλαιακών απαιτήσεων, καλύτερη πρόσβαση στην αγορά, διαδικασίες εξυγίανσης και με τον τρόπο αυτό προκύπτουν ε, τράπεζες που είναι πολύ πιο ανθεκτικές. Αυτό λοιπόν ε, που δείχνουμε στις αναλύσεις μας και στα business model, το δείξαμε πριν από κάποια χρόνια, είναι ότι οι τράπεζες ε, ε, ήταν πολύ πιο αποτελεσματικές όταν άλεξαν τα υποδείγματά τους, όταν εντόπισαν τους ε, τομείς ε, που αποφέρουν κέρδη, τους προέβαλαν αυτούς τους τομείς και άφησαν άλλους που δεν ήταν κερδοφόροι. Επίσης, οι τράπεζες που επένδυσαν στη νέα τεχνολογία κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν τη μετάβαση και να είναι πλέον σε πολύ πιο σταθερή εξέλιξη. να κάνω μια δεύτερη ερώτηση γιατί έχω χρόνο ακόμα που μοναλογεί, ε, ασκείται κριτική για το γεγονός ότι ομολογίουχοι αγοράζουν πολλά ομόλογα της δικής τους της ε, τράπεζες. Άρα η έκθεσή τους είναι πολύ υψηλή. Το 2018 μάλιστα αυξήθηκε αυτή η έκθεση στην Ιταλία και την Πορτογαλία και αυξήθηκαν και οι αποδόσεις κινδύνου. Τι σκέφτεστε να κάνετε για να ανακόψετε αυτή την τάση. Νομίζω ότι το ανέφερα αυτό στην απάντηση που έδωσα στον ε, κύριο Γκαρικάνο. Πράγματι έχουμε εργαλεία στην εργαλειοθήκη μας για να αντιμετωπίσουμε τα ανοίγματα σε κρατικά ομόλογα. Ε, κάνουμε τεστ τα οποία βεβαίως ε, αφορούν τις τράπεζες και κατόπιν οι τράπεζες είναι εκείνες, αλλά και εμείς, μάλλον εμείς είμαστε εκείνοι που ορίζουμε το ανάχωμα που πρέπει να υπάρχει, το απόθεμα στις τράπεζες για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι. Ε, τώρα, όσον αφορά τους κινδύνους ε, και τους ομολογιούχους, εκεί γίνονται τεστ στον πυλώνα 2 και εκεί μπορούμε βεβαίως ε, να εκθέσουμε και συγκεκριμένες ε, συμβουλές. Αυτό κάνουμε με τα στρες για τους ομολογιούχους. Γκούμπαρ εκ της Θα μιλήσω πορτογαλικά. Δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη έχει να κάνει με το ότι εμείς εργαζόμαστε με μια οικονομική πολιτική συντονισμένη. Όμως υπάρχει μεγάλη δυναμία, οπότε εγώ ρωτάω, μπορούμε να συνεχίσουμε να επιμένουμε στις προσπάθειες αυτές για να ξεπεράσουμε τον εθνικό κατακαιρματισμό που υπάρχει στο χρηματοπιστωτικό τομέα πανευρωπαϊκά. Υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση ευρωπαϊκών τραπεζών υπάρχουν οι μεγάλες και μία από τις διαγνώσεις που έχουν γίνει με την τελευταία χρηματοπιστωτική κρίση είναι ότι οι μεγάλες τράπεζες είναι πολύ γερές μέχρι που να πάψουν να είναι. Τώρα το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στο θέμα των εγγύσεων καταθέσεων και η Τραπεζική Ένωση τελικά καταλήγει να κουτσένει. Και τι θα γίνει με όλα αυτά τα οποία μένουν μόνο στα χαρτιά και δεν εφαρμόζονται. Από την άλλη, βλέπουμε να υπάρχουν παρεμβάσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Κομισιόν. Δεν ξέρουμε τελικά ποιο είναι αυτό που διευθύνει όλε αυτέ τι διαδικασίε. Και εξαρτάται κάθε φορά από την πολιτική δύναμη που διαθέτει ο κάθε υπεύθυνο ή κάθε χώρα. φοβάμαι πως τελικά είναι οι φορολογούμενοι οι οποίοι πληρώνουν την ύφη. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω κατά πόσο εσείς θεωρείτε ότι το πρόβλημα αυτό, το ότι ο έλεγχος και η υπευθυνότητα δεν συνδέονται, αν πιστεύετε ότι λύνεται με περισσότερη κεντρική προσέγγιση ή μήπω αντίθετα μπορεί να λυθεί καλύτερα με την αρχή αυτή που λέει ότι όποιος πληρώνει αποφασίζει τελικά. Uh, Σας ευχαριστώ. Ίσως τα έχετε ήδη ακούσει από μένα, αλλά θα τα ξαναπώ. Όσον αφορά το θέμα της συγκέντρωσης ή το θέμα του εθνικού κατακαιρματισμού, πολύ μεγάλη μια τράπεζα για να χρεοκοπήσει. Κοιτάξτε, στο αμερικανικό σύστημα είδατε πώς αντιμετωπίστηκε η κρίση. Και υπάρχουν κοινά σημεία ανάμεσα στο Πορτορίκο και την Ελλάδα. Δύο χώρε, τέλο πάντων μια πολιτεία και μια χώρα, ίδιου μεγέθου λίγο πολύ, που είχαν πρόβλημα με το κρατικό χρέο. Και οι τράπεζε στι χώρε αυτέ βρέθηκαν φυσικά σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Στο Πορτορίκο είχατε τι τράπεζε, οι οποίε έκλεισαν πριν το Σαββατοκύριακο, μετά υπήρξε η διάσωσή τους και βοήθησαν τράπεζες από άλλες πολιτείες. Ο κίνδυνος δηλαδή του τραπεζικού τομέα σε μια πολιτεία απορροφήθηκαν με την παρέμβαση τραπεζών από άλλη πολιτεία. Κάτι το οποίο βοήθησε ήταν ένας επιμερισμός κατά κάποιο τρόπο. Και μειώθηκε η ανάγκη παρέμβασης ε, των κρατικών αρχών της κυβέρνησης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα, έχουμε έναν φαυλοκύκλο μεταξύ τραπεζών και κρατικού χρέους που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Και ακόμα οι ελληνικές τράπεζες έχουν πολύ ψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οπότε το βασικό θέμα είναι ότι πρέπει να χτίσουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι πιο γερό και ο τραπεζικός ε, κλάδος να μπορεί να παίξει ρόλο επιμερισμού κινδύνου αντί να αμβλύνει ε, αντί να, να μεγαλώνει τους κινδύνους. Ένα τέτοιος μηχανισμός χρειάζεται και είναι σημαντικό να συμφιλιώσουμε, όπως λέτε, ε, τους ελέγχους με το δίκτυο ασφάλειας. Εγώ δεν θα πήγαινα πάντως τόσο μακριά ώστε να πω ότι υπάρχει παρέμβαση από τις ευρωπαϊκές αρχές. Όχι. Υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο που διέπει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχει συγκεκριμένες ευθύνε και αρμοδιότητες για τις τράπεζες όλες τις χώρες ε, μέλη που συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση. Οπότε δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο αυτή η παρέμβαση εδώ. Ευχαριστούμε δεύτερο ο γύρο. Αλλά τέσσερα λεπτά τώρα και θα είμαι και αυστηρό, γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Καρβέρτ Κρίστους από κύριο Κίρτσο. Ε, το μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το ύψος των ε, μη εξυπηρετούμενων οφειλών, non-performing loans, το οποίο δημιουργεί, είναι ρεκόρ βέβαια στην Ευρωζώνη και δημιουργεί προβλήματα στις τράπεζες αλλά και στην οικονομία. Υπάρχει μία, σύμφωνα ε, με, το, με τις οικονομικές σελίδες του ελληνικού τύπου, το οικονομικό ρεπορτάζ, υπάρχει μια πρόταση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ε, που στηρίζεται σε αυτά που έγιναν και στην Ιταλία το 2018 και με βάση αυτή την πρόταση, την οποία προωθεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, ε, non-performing loans, κόκκινα δάνεια, ίσως άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα περάσουν ε, από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες σε ένα σχήμα προστασίας ενεργητικού Asset Protection Scheme, APS, και αυτό το σχέδιο αναμένεται να, ε, να πραγματοποιηθεί, δηλαδή να ξεκινήσει η εφαρμογή του το, στα τέλη του 2019. Ε, θα ήθελα την άποψή σας, δηλαδή πώς ακριβώς ε, πρέπει να διαχειριστούμε το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, και βέβαια ήθελα και την άποψή σας για τη διαφορά στο επιτόκιο. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι το επιτόκιο στα δάνεια μέχρι 250.000 στην Ελλάδα, το μέσο επιτόκιο, είναι 4,9%, όταν το μέσο επιτόκιο στην Ευρωζώνη για τα ίδια δάνεια μέχρι 250.000 είναι 2,06%. Δηλαδή έχουμε 2,5 φορές υψηλότερο επιτόκιο στην Ελλάδα, ε, ενώ χρειαζόμαστε ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Ε, ποια είναι η άποψή σας, γιατί πρέπει να σας πω ότι η ελληνική κοινή γνώμη στηρίζει πολλά σε εσάς. Ευχαριστώ. Well, thank you very much. Uh, first of all, let me say that... Uh, Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θέλω να πω ότι οι ελληνικέ τράπεζε είναι ιδιαίτερα δραστήριε σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έχουν καταφέρει να επιτύχουν το στόχο που συμφωνήσαμε με τι τράπεζε τα περασμένα χρόνια. Πολύ σωστά ε, αναφέρεται ότι παραμένει, πολύ ψηλά κάποια επίπεδα και είναι 41% ε, το μέσο επίπεδο. Χρειαζόμαστε λοιπόν περαιτέρω πρόοδο. Έχουν, έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους, αλλά ακόμη και αν επιτύχουν ε, τους φιλόδοξους στόχους, μείωση κατά δύο τρίτα ε, των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα παραμείνει ένα 18% στο τέλος της διαδικασίας. Ε, όπως σας έχω πει πολλές φορές λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται και περαιτέρω πρωτοβουλίες. Κατά τη γνώμη μου η πρόταση ε, του Ελληνικού ε, Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που υποστηρίζεται από την ελληνική κυβέρνηση είναι καλή πρόταση. Έγινε και μια πρόταση από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστεύω και νομίζω ότι στην παρούσα συγκυρία αν θέλεις να αντιμετωπίσεις ένα τόσο μαζικό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων χρειάζεται ένα εργαλείο, ε, κάποια μορφή εργαλείων στην Ιταλία έχουν λειτουργήσει οι εγγυήσει τυκλοποίηση, μειώσαν ε, τον όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πιστεύω λοιπόν ότι και στο ελληνικό πλαίσιο θα υπάρξει ε, βελτίωση και συνεργαζόμαστε στενά και με τις τράπεζες και με τις αρχές στην Ελλάδα προς το σκοπό αυτό. Για τα επιτόκια και πάλι είναι σαφές ότι αν οι τράπεζες έχουν υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων, αν το περιβάλλον κινδύνου είναι πολύ ε, ε, ευάλωτο. Αυτό αποτυπώνεται και στις τιμές. Είναι περισσότερο θέμα αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών γενικότερο παρά να έχουμε παρεμβάσει στα επιτόκια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μαργαρίτα Μάρκες εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Έχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν να μειώσουν τους κινδύνους στον τραπεζικό τομέα. Πρέπει να συνεχίσουμε να μειώνουμε τον κίνδυνο στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, το παρόν επίπεδο σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι πολύ υψηλό στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα πρέπει να γίνεται παράλληλα με τη δημιουργία μιας δευτερογενου αγοράς για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η πρώτη ερώτησή μου είναι η εξή. Πιστεύετε ότι η ΕΚΤ μπορεί να συνεισφέρει στην περαιτέρω εμβάθυνση τη δεύτερογενού αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δεύτερη ερώτηση. Έχουν εφαρμοστεί σχέδια δράσης με αρκετή επιτυχία, προσπαθώντας να διασφαλίσουν ότι και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο θα μπορέσουν να βελτιωθούν τα ε, πλαίσια ε, για την πτώχευση και θέλουμε να έχουμε ένα σαφέστερο και πιο προβλέψιμο πλαίσιο σύμφωνα με αυτά που είπατε και εσείς όταν είχατε εκλεγεί στον τωρινό σας ρόλο, που είχατε πει ότι δεσμεύεστε υπέρ της διαφάνειας. Πρέπει λοιπόν τα πλαίσια να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση η διαφάνεια να μην παραμένει στα λόγια, αλλά να κατευθύνουμε τις δραστηριότητες ε, δημοσιοποίησης προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τραπεζών για να βελτιώσουμε την ε, πειθαρχία στην αγορά με στόχο την καλύτερη εποπτεία και καλύτερο έλεγχο των κινδύνων που αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Η τρίτη μου ερώτηση. Το Δεκέμβριο του 2018 ζητήθηκε από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτευχθεί πρόοδος στην Ένωση Τραπεζών. Συμφώνησαν να υπάρχει ως μηχανισμός ασφαλείας ε, ένα ταμείο εξυγίανσης που όμως δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι ότου να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Ο τρίτος πυλώνας της Ένωσης Τραπεζών η ερώτησή μου είναι, θα αναλάβετε ενεργά ε, μέτρα ώστε να πείσετε αυτούς που μέχρι τώρα έχουν μπλοκάρει αυτό το μηχανισμό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, on your point on the... Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, όσον αφορά την μείωση, το ενδεχόμενο μείωση σε το μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη δευτερογενή αγορά, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω, όπω υπενήχθηκα και προηγουμένω στην απάντηση που έδωσα, ότι η πρόοδο είναι πολύ σημαντική και ε, για να είμαι ειλικρινή, η δεύτερογενή αγορά λειτουργήσε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Ε, μερικοί από εσά θα θυμάστε ότι πριν από δυόμιση χρόνια πρότεινα να υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια, ένα κεφαλαίων ακριβώς ε, διότι θεωρούσα ότι η δευτερογενής αγορά δεν ήταν αρκετά έτοιμη για να αντιμετωπίσει το θέμα. Πρέπει όμως να πω ότι εξελίξει στη ρευστότητα της αγοράς, αλλά και πάρα πολλές υπηρεσίες που προσφέρονται, όλα αυτά αυξήθηκαν σημαντικά. Η ΕΚΤ Βεβαίω, και υπήρξαν ε, πρωτοβουλίες από εμάς και από την ΕΚΤ ε, για να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και η ΕΚΤ ε, έχει δρομολογήσει πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα ένα είδος ε, eBay, ένα είδος ε, εισόδου πύλης, μία πύλη με συγχωρείτε, εισόδου ε, για αυτούς που ενδιαφέρονται ενδεχομένως. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου. Κατά τα άλλα, όσον αφορά το καθεστώς ε, πτώχευσης, ε, το benchmarking, ε, την διαφάνεια στις προβλέψεις, κοιτάξτε, προβλεψιμότητα και διαφάνεια, αυτά τα έχουμε βελτιώσει. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε την πολιτική μας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αυτό είναι ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Δημοσιεύουμε πάρα πολλές από τις μεθόδους μας, προγραμματίζουμε να δίδουμε περισσότερες πληροφορίες, να προχωρεί το ενδεχόμενο της συγκρίση χρησιμότητας. Πράγματι και εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και πειθαρχία στην αγορά. Ε, νομίζω ότι όσον αφορά την ΕΚΤ, η έκτα έχει ήδη τοποθετηθεί έχει ε, τοποθετηθεί στο ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε αυτό τον τομέα και πράγματι θέλουν να στηρίξουν και την περαιτέρω πρόοδο. Επόμενος ερωτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα ήδη στην αρχή ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συζητήθηκαν σήμερα αρκετά. Και στην Ιρλανδία τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και οι τράπεζες από 15% το 16 έφτασαν τώρα στο 4 περίπου Άρα δηλαδή τεράστια η πρόοδος των Ιρλανδικών τραπεζών να βγάλουν τα κόκκινα δάνεια από τους ε, ισολογισμούς τους. Οι τράπεζες της Ιρλανδίας βέβαια χρεώνουν διπλάσια επιτόκια από το μέσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δανεισμό ε, στις επιχειρήσεις. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι η Ιρλανδική οικονομία αυξάνεται ταχύτατα, όμως ε, η η κίνδυνοι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά τον Brexit είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ως εκ τούτου θέλω να ρωτήσω πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των υψηλών επιτοκίων στην Ιρλανδική οικονομία λόγω του γεγονότος ότι η και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες ε, είναι πλήρως και πολύ σωστά ανεξάρτητες από τις κυβερνήσεις. Όμως αυτό το συγκεκριμένο θέμα πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε τη στιγμή που υπάρχει μια συστημική προσέγγιση των τραπεζών να αποκομίζουν κέρδη επιβάλλοντας υπερβολικά επιτόκια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις υποθήκες. Άρα δηλαδή τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τώρα δεν είναι δικαιολογία πια στην Ιρλανδία. Τώρα, όσον αφορά το Brexit, μήπω έχετε κάνει κάποια ανάλυση, όχι όσον αφορά τι ε, τράπεζε που θα έρθουν στην Ευρωζώνη, αλλά το θέμα του κινδύνου που μπορεί να προκύψει για οικονομίε, οικονομίε που θα εκτεθούν σε αποχώρηση χωρί συμφωνία. Το θέμα τη ε, ισοτιμίας ανάμεσα στη Στερλίνα και την Ευρωζώνη. Αυτά τα δύο θέματα. Πού ακριβώ βλέπετε τον εποπτικό σα ρόλο, πρώτον όσον αφορά το επιτόκια και δεύτερον να διασφαλίσετε ότι θα υπάρχει ένας μηχανισμός ε, για τα κρατικά χρέη και για τις τράπεζες στην περίπτωση που θα έχουμε το Brexit. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. σε σχέση με αυτό που είπατε για ότι υπάρχει σημαντική πρόοδο των Ιρλανδικών τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ θετικά. Όσον αφορά το επιτόκιο ε, που αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σχόλιο. Αν δείτε τις προηγούμενες ε, κρίσεις, θα δείτε ότι υπάρχει ένας πιστοτικός κύκλος που σε ορισμένου τομεί οδηγούσε προς μια φούσκα ε, και υπήρχαν και υπερβολικά επιτόκια και υπερβολική χορήγηση πιστώσεων. Το σύστημα λοιπόν το οποίο εδραιώθηκε σημαίνει ότι οι εθνικές αρχές και μακροπροληπτικά μπορούν να αρχίσουν να εφαρμόζουν μακροπροληπτικά εργαλεία όταν βλέπουν υπερθέρμανση σε κάποιους τομείς. Αν δείτε λοιπόν στον τομέα των ακινήτων ότι υπάρχει ε, δημιουργία μιας φούσκας, Μπορείτε να δείτε το λόγο προς την τιμή των ακινήτων κλπ. για να έχετε κάποια προστατευτικά μέτρα. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από διάφορα κράτη-μέλη ε, στον κύκλο των πιστώσεων δημιουργούν κάποια επίπτωση και στον κύκλο των επιτοκίων. Τώρα, για το άλλο που ρωτήσατε, όπως έλεγα και πριν, θα πρέπει να υπάρχει πειθαρχία ε, και ανταγωνισμός. Δηλαδή θέλετε οι τράπεζε να είναι ικανέ να μπαίνουν στα αγορά. Αν σε ορισμένε δικαιοδοσίες υπάρχουν υπερβολικά επιτόκια, ο ανταγωνισμός αναμένεται να εξισορροπήσει κάπως την κατάσταση. Η ολοκλήρωση των αγορών δυστυχώς δεν είναι ακόμη σε τέτοιο επίπεδο που να επιφέρει αυτές τις θετικές εξελίξεις. Όσον αφορά το Brexit, βεβαίως και μελετούμε πολύ προσεκτικά τις επιπτώσεις επί των τραπεζών, όχι μόνο για ε, ε, το που βρίσκονται, αλλά και για την έκθεση των ε, τραπεζών. Και οι συνάδελφοι από τον τομέα της σταθερότητας στην ΕΚΤ εξετάζουν αυτό το θέμα. Αν το δείτε στατικά, αν κάνετε μια στατική αξιολόγηση, το συμπέρασμα είναι ότι είναι διαχειρίσιμος ο κίνδυνος. Ναι, αν συνδυάσει βέβαια κανείς το μακροοικονομικό σοκ, τις ενοχλήσεις στο εμπόριο, τις μετατοπίσεις εταιριών, σαφώς πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση εξετάζοντας τους πιθανούς κινδύνους. Ευχαριστώ πολύ. Και τελευταί... τελευταίος ομιλητής από το ΕΛΚ, Στέφαν Μπέργκερ. Uh, το ερώτημα μου αφορά τα κρυπτονομίσματα συγκεκριμένα την επόμενη χρονιά εμφανίστηκε, θα εμφανιστεί από το facebook το Libra. Πολλοί έχουν λάβει προειδοποίηση για αυτό το θέμα. Η ε, καταναλωτές ε, θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από το ευρώ και το Λίμπρα θα μπορούσε να είναι ένα πρόβλημα ε, για την κεντρική τράπεζα. Αυτό δημιουργεί πολλές ανησυχίες, ξέπλυμα βρωμικού χρήματος, τρομοκρατία και πολλά άλλα. Η ΕΚΤ θα πρέπει να αντιμετωπίζει το Λίμπρα ως ένα καμπανάκι κινδύνου και ερωτώ θα μπορούσε να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σταθερό νόμισμα που να εκδίδεται, να στηρίζεται από την ΕΚΤ ή να υπάρχει ε, κάποια εναλλακτική λύση, γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει τέτοιου είδους εναλλακτική λύση στην ε, Ευρωζώνη. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ε, ο προτινόμενος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ έκανε μία ομιλία προχθές και εκεί έθιξε πολλά από τα θέματα που αναφέρετε. Θέλω να σας πω από πλευράς ε, εποπτείας. Εμένα αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα είναι η συμβατότητα με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Ε, παλαιότερα κάναμε μία ανάλυση για τους κινδύνους που συνεπάγονται τα κρυπτονομίσματα. Ε, το σημαντικότερο είναι ε, θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα. Αυτό είναι μία απόλυτη προϋπόθεση. Μέχρι τώρα, όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, οι πελάτες ε, πρέπει να είναι ενημερωμένοι ότι αν επενδύσουν χρήματα σε τέτοιους ε, κρυπτονομίσματα κινδυνεύουν να χάσουν όλα τους τα χρήματα. Τους προειδοποιούμε, αλλά δεν μπορούμε να λάβουμε την πλήρη ευθύνη. Εμείς τους προειδοποιούμε ότι δεν υπάρχει δίχτυα ασφαλείας για τέτοιου είδους νομίσματα. Βεβαίως, ε, αν υπάρχει τώρα μια λειτουργία, μια, ένα φαινόμενο όπως αυτό με το Libra και αυτό επεκταθεί τα μάλα, θα πρέπει να αναθερήσουμε ίσως και εμείς τη στάση μας. Αυτή τη στιγμή γίνεται αρκετή δουλειά και σε επίπεδο G7 ε, και στο ε, μηχανισμό σταθερότητας. Ε, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία και πράγματι η απάντηση θα πρέπει να δοθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Τελευταίος, Φαρνάντες. S&D, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνα με το σχέδιο του Δεκεμβρίου του 2018 για την καταπολέμηση της νομοποίησης παράνομων εσόδων, τέθηκε το θέμα της τιτλοποίησης. Ε, είπαμε ότι πρέπει να διευκρινιστεί ο βαθμός στον οποίο θα γίνεται με την άδεια των αρχών όταν έχουν επαληφθεί οι κανόνες EML και SFT. Έπειτα πρέπει να υπάρχει μια εμοιόμορφη ερμηνεία της γλώσσας η οποία χρησιμοποιείται για τους κανόνες αυτούς, ML και SFT. Τρίτον, πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια και να μπορούν να δράσουν οι μακροπροληπτικές αρχές ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιους κινδύνους πάντα βάσει των κανόνων EML και SFT. Μπορείτε λοιπόν να μας ενημερώσετε τι δουλειά γίνεται και πόσο, πώς προχωράει αυτή η υπόθεση. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ε, συγγνώμη που σας στέλνω πίσω το μπαλάκι, αλλά βλέπετε χρειάζεται νομοθετική δράση για να προχωρήσουν όλα αυτά. Το θέμα της ε, αδειοδότησης, πώς δηλαδή θα παίρνουμε πίσω μια άδεια, θα φερούμε μια άδεια. Σε μερικές περιπτώσεις έχετε μια μεγάλη ανησυχία για μια τράπεζα που μπορεί να κινδυνεύει να χρεοκοπήσει, αλλά τότε στην εθνική νομοθεσία δεν έχετε τα εργαλεία τα απαραίτητα έτσι ώστε να μπει στη διαδικασία χροκοπίας η τράπεζα και είναι δύσκολο να ξεκινήσει μια διαδικασία αφαίρεση της άδεια. Χρειάζεται λοιπόν αναρμόνιση του νομικού πλαισίου, ώστε όταν υπάρχουν τέτοιε περιπτώσει να υπάρχει μια ισχυρή νομική βάση, ώστε να μπορούμε να αφαιρέσουμε την άδεια αμέσω. Όσον αφορά τώρα του τραπεζικού κλάδου, τις ε, θηγατρικές μάλλον. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι για τις θηγατρικές αυτός είναι τομέας ε, την ε, αρμοδιότητα του οποίου έχει χώρα στην οποία βρίσκεται η τράπεζα. Ακόμα και αν είναι μια εστονική ή μια δεν ξέρω τι, υπάρχουν προβλέψεις για την συνεργασία. Σε ένα βαθμό το ML5 τα έχει ρυθμίσει αυτά, αλλά όντως χρειάζεται ένα ισχυρό πλαίσιο. Δεν θέλουμε μέλες ευτή ε, επόπτη. Χρειάζεται ενίσχυση της συνεργασίας των εποπτικών αρχών, των δικών μας ε, δηλαδή, και των αρμοδίων αρχών στις χώρες μέλη. Σίγουρα επιδέχεται βελτίωση το θέμα των θηγατρικών. Ξέρετε ότι αν πρόκειται για θεατρική τρίτης χώρας, δεν είναι τότε ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά των εθνικών αρχών. Οπότε το πώς αντιμετωπίζει κανείς αυτές τις περιπτώσεις είναι πιο περίπλοκο. Όντως επιδέχεται πρόοδο το θέμα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ολοκληρώνεται αυτό το τμήμα της συνεδριάσεώς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ανδρέα Ενρία που ήταν μαζί μα και που μα αφιέρωσε τόσο χρόνο και προσπάθεια για να απαντήσει στις ερωτήσει μα. Και εσάς σας ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε του χρόνου σα. Έχουμε 10 λεπτά για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, το οποίο θα είναι πολύ εντατικό. Αλλά να ξεκινήσουμε ακριβώς στις 10.30. Ευχαριστώ. Και νομίζω το Δεκέμβριο θα τον ξανά έχουμε τον κύριο Ενρία μαζί μας για να συνεχίσουμε.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 Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αρχίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερες ερωτήσεις. Καθίστε λοιπόν παρακαλώ και παρακαλώ και τον τύπο, τους φωτογράφους να μας επιτρέψουν να αρχίσουμε. Thank you. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε στο σημείο 5 της ημερήσιας ε, διάταξης και πάλι ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του κύριου Γκουλτιέρη, του Πρόεδρου μας που δεν μπορεί να είναι εδώ, οπότε αναλαμβάνω εγώ να προεδρεύσω αυτή τη τόσο σημαντική συνεδρίασης. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που μπορώ να καλωσορίσω εδώ την κυρία Κριστίν Λαγκάρτ που είναι υποψήφια για τη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως γνωρίζουμε, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Επιτροπής, ο τωρινός ο κύριος Δράγκη, αποχωρεί την 31η Οκτωβρίου μετά από πέντε χρόνια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 283 σημείο 2 τη ε, συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί μετά από σύσταση του Συμβουλίου για τον ορισμό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα έχουμε αυτήν την ε, δημόσιο ακρόαση. Προηγουμένως ε, υποβλήθηκαν γραπτά 176 76 ερωτήσεις και θα βρείτε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις της κυρίας Λαγκάρτα στο σφακέλου σας. Στις 6 θα ψηφίσουμε σήμερα και μετά θα υποβάλουμε πρόταση προς απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη σύσταση του Συμβουλίου για τον ορισμό της κυρίας Λαγκάρτα στη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στην σύνοδό του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 16 με 19 Σεπτεμβρίου θα ε, ψηφίσει επ' αυτού. Θα ακούσουμε για 10 λεπτά την κυρία Λαγκάρτ και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Έχουμε ένα τεράστιο κατάλογο ευρωβουλευτών που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις, οπότε εγώ θέλω να προσπαθήσω να προλάβουμε να έχουμε και λίγο χρόνο για το catch the eye στο τέλος. Οπότε ζητώ στην κυρία Λαγκάρτ να τηρήσει το χρόνο της, όπως και εσείς βέβαια, και να είσαστε ρεαλιστές. Αν πιστεύετε ότι με την ερώτησή σας μπορείτε να έχετε και κάποιες ουσιώδεις απαντήσεις, ε, κάντε την. Λοιπόν, 10 λεπτά καταρχήν η κυρία Λαγκάρτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θα αρχίσω ε, ζητώντα ε, κάποια πήκη από εσά. Γιατί εγώ είχα ετοιμάσει 15 λεπτά παρέμβαση. Το συζήτησα χθε με τον κύριο Γκουαλτιέρη και νόμιζα ότι είχα 15 λεπτά στη διάθεσή μου. Αλλά αν πρέπει να σταματήσω στα 10, θα σταματήσω στα 10. Κανένα πρόβλημα. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ στην ε, Επιτροπή σας. Και ομολογώ ότι αισθάνομαι και κάπως ε, περίεργα συναισθαλμένα εδώ, γιατί Πολλοί από εσά έχουν βρεθεί κάποια φορά στην δικιά μου θέση. Δηλαδή είσαστε υποψήφοι για κάποια θέση, σιγά σιγά μαθαίνετε και σιγά σιγά αποκτάτε τον ε, ενθουσιασμό που χρειάζεται για να εξυπηρετήσετε το σκοπό σας. Πιστεύω ότι οι σχέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Νομισματικής Ένωσης. Η κεντρικοί τραπεζίτέ είναι ανεξάρτητοι. Δεν εκλέγονται όμως απευθεία από το κόσμο. Οπότε λογοδοτούν μόνο σε αυτούς οι οποίοι εκλέγονται άμεσα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως αποτελεί ένα στοιχείο κλειδί στον ορισμό μου. Σήμερα το πρωί δίστασα αν ήθελα να σας παρουσιάσω την ευρωπαϊκή οικονομική κατάσταση, να σας δώσω μια τεχνική κατάσταση για την νομισματική πολιτική. Και αποφάσισα ότι είναι ίσως πιο ενδιαφέρον να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στην επαγγελματική μου εμπειρία και το υπόβαθρο που έχω και που σχετίζεται με τα καθήκοντά μου εφόσον αναλάβω την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ήμουν λοιπόν επικεφαλής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα τελευταία 8 χρόνια και είχα το προνόμιο να είμαι επικεφαλής ενός οργάνου που βρίσκεται στην καρδιά της οικονομικής ασφάλειας ε, στον κόσμο και συνεργάζεται με τις ε, κεντρικές τράπεζες. Επίσης ήμουν υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας και τότε συνέφερα στην επίλυση κρίσεων με εργαλεία, με ρυθμίσεις τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, έχω συμμετάσχει στην ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Τώρα, τι είναι αυτό το οποίο με οδήγησε να αναλάβω τα καθήκοντα αυτά. Πρώτα απ' όλα ήμουνα αποφασισμένη και πίστευα και πιστεύω ακόμα ότι είναι πολύ σημαντικό να προσφέρει κανείς στο κοινό και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του κόσμου. Δυστυχώς έμαθα τις αρνητικές επιπτώσεις της έλλειψης ρυθμίσεων ή της έλλειψης αποφάσεων και πόσο αρνητικά επηρεάζουν το κόσμο. Και κατάλαβα ότι οι αποφάσεις των ε, θεσμών επηρεάζουν πάρα πολύ τις ζωές του κόσμου. Από τις θέσεις που κατήχα κατά το παρελθόν, πάντα πίστευα ότι οι αποφάσεις αυτές είναι κάτι πολύ σημαντικό. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσπαθήσαμε να επικεντρωθούμε και στην ε, μείωση των ανισοτήτων, ε, να προστατεύσουμε ε, το περιβάλλον από την κλιματική αλλαγή, να φροντίσουμε για μια ανάπτυξη με τη συμμετοχή όλων. Αυτά όλα μπορεί να μην θεωρούνται τα κύρια καθήκοντα που είναι μακροοικονομική πολιτική. Όμως τελικά πιστεύω ότι θεωρούνται και μακροοικονομικά στοιχεία σήμερα. Μια καλή ηγεσία δεν σημαίνει μόνο ότι θέτουμε προτεραιότητες, σημαίνει επίσης ότι ακούμε και ακούμε όλες τις ε, φωνές, όχι μόνο των εμπειρογνωμόνων, των ειδικών, αλλά όλων. Και επίσης βασιζόμαστε και στη διαφοροποίηση της σκέψης. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνεργάστηκα στενά με σημαντικούς οικονομολόγους. Προκειμένου να μας δίνουν στοιχεία που βασίζονται σε δεδομένα και άκουσα πάντα προσωπικά και το προσωπικό, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια σύγχρονη προσέγγιση του έργου μας, προκειμένου να συμμετέχουν περισσότερο όλοι στο έργο του Διεθνούς Μασνατικού Τομείου και να βοηθήσουμε την κοινωνία. Αυτή ήταν η στρατηγική μου. Και γιατί συνεχίζει να είναι, γιατί ακριβώ αυτές οι ίδιες ε, αξίες είναι στις οποίες εξακολουθώ να πιστεύω και θα προωθήσω εφόσον τελικά επικυρωθεί η θέση μου στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλω να αναφερθώ σε τρεις αρχές που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές στο μελλοντικό μου έργο. Οι πρώτες ε, δύο που θα εξετάσω μαζί είναι η δέσμευση υπέρ της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζης. Η δεύτερη είναι η ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Αυτά τα δύο θα τα συζητήσω μαζί σας μαζί. Και το τρίτο είναι η συμμετοχή όλων. Να μην υπάρχουν αποκλεισμοί δηλαδή. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Λοιπόν, δέσμευση και ευελιξία. Γνωρίζουμε και το γνωρίζουμε από δεκαετίας θεωρίας και πράξης ότι μια σαφής εντολή για την νομισματική πολιτική είναι πολύ βασική, όπως επίσης και η δέσμευση της Κεντρικής Τράπεζας να πετύχει τους στόχους της. Και αυτό το έχει δείξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την αρχή. Τα πρώτα χρόνια πέτυχε να ηγηθεί μιας ε, νομισματικής ένωσης με πάρα πολλές ε, διαφορές, κρατώντας ε, χαμηλά και σταθερό τον πληθωρισμό. Και μετά φτάσαμε το 2008 που έπρεπε να αντιμετωπίσει όχι τον πληθωρισμό αλλά τον αποπληθωρισμό. Και πάλι όμως η δέσμευσή της και η αποφασιστικότητά της ήταν ζωτική σημασία προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των τιμών σε μια περίοδο χαμηλού πληθωρισμού. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσαρμόστηκε στις νέες προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει. Οπότε ξεπέρασε τις παλιές πεπιθήσεις με τις νέες εμπειρίες και ήταν καινοτόμο στην πολιτική της με τη νέα της εργαλειοθήκη στα πλαίσια βέβαια πάντα που θέτει ο νόμος και η εντολή της. Και ακριβώς αυτή, αυτή η προσαρμοστικότητα, αυτή η ευελιξία που απέδειξε ότι διαθέτει βοήθησε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες συνθήκες. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα καινοτομία και προσαρμογής, σίγουρα η κρίση, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των περισσότερων εμπειρογνωμόνων, θα ήταν πολύ χειρότερη. Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε επίση κάποιε έρευνε για να εκτιμήσει τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε υπάρξει αυτή η καινοτομία, αν δεν είχε αντιμετωπίσει με προσαρμοστικότητα την κρίση. Ε, λοιπόν η οικονομία θα ήταν κατά 2% σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι τελικά. Αν, δίχα, αν δεν είχε ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από το 2014 μη συμβατικά μέτρα. Ήταν πολύ σημαντικό που ελήφθησαν και τέτοια μέτρα. Η απασχόληση επίσης βελτιώθηκε κατά 11 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια νέες Θέσει απασχόληση μετά από τα μέσα του 2013, γιατί ακριβώ αυτά τα μη συμβατικά μέτρα δημιούργησαν και πάλι εμπιστοσύνη στον κόσμο. Εφόσον επιβεβαιωθεί η θέση μου επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λοιπόν, θα ακολουθήσω αυτέ τι αρχέ. Την ε, δέσμευση αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για προσμαστικότητα, για ευελιξία ε, σε σχέση με τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται γύρω μας. Η προκλήσεις που αντιμετώπισε βέβαια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχουν εξαφανιστεί. Η Ευρωζώνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κινδύνους που έχουν να κάνουν κυρίως με εξωτερικούς παράγοντες και ο πληθωρισμός παραμένει, εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός και σίγουρα πιο χαμηλός από το στόχο. Συμφωνώ λοιπόν με την άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι χρειάζεται μία πολιτική προσφοράς χρήματος προκειμένου ο πληθωρισμός να επιστρέψει στο περίφημο κάτω αλλά κοντά στο 2%. Όμως υπάρχουν και μερικά σημαντικά ζητήματα που έχουμε μπροστά μας και που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η νομισματική πολιτική. Πρώτα απ' όλα, ότι οι επιπτώσεις των μη συμβατικών πολιτικών να εξακολουθούν να είναι θετικές και για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τι αρνητικέ παρενέργειε, για τις παρενέργειες που μπορεί να προκληθούν από τέτοιες πολιτικές και να λάβουμε υπόψη μας και τι ανησυχίε του κόσμου. Παραμένουμε λοιπόν δεσμευμένοι στην εντολή μας που είναι για σταθερότητα τιμών, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση ε, κόστου και ωφέλου. Δεύτερον, το περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού και χαμηλών επιτοκίων επίση θέτει ερωτήματα στρατηγική για όλε τι κεντρικέ τράπεζε, όχι μόνο την Ευρωπαϊκή. Οι κεντρικέ τράπεζε λοιπόν πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα ποια είναι η δυναμική του πληθωρισμού και να χρησιμοποιήσουν νέα μέσα τα οποία μπορούν να περιορίσουν την κρίση και να χρησιμοποιήσουν ε, ισολογισμού και μη συμβατικέ πολιτικές. Και πρέπει επίση να προβληματιστούν για το κατά πόσο τα δικά του νομισματικά πλαίσια πολιτική είναι επαρκή για να αντιμετωπίσουν μελλοντικέ προκλήσεις. Και αυτό είναι ένας στόχο που εγώ θα αναλάβω εφόσον ε, αναλάβω επικεφαλής της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζας. Τρίτον, οι κεντρικέ τράπεζε όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουν νέα είδη προκλήσεων. Κλιματική αλλαγή, ε, τεχνολογικές αλλαγές, ε, κατακαιρματισμός της πολυμερούς τάξης που έχουμε σήμερα στον κόσμο. Και είναι πολύ σημαντικό η νομισματική πολιτική να βλέπει μακριά και να λαμβάνει υπόψη της το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να πετύχει τη σταθερότητα των τιμών, που είναι και εντολή της. Τέλος, η αποτελεσματικότητα της νομισματικής μας πολιτικής έχει να κάνει με την αντοχή του ε, χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ρόλος της όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχει ενισχυθεί, τη ζητήθηκε να αναλάβει νέες αρμοδιότητες για μακροπροληπτική πολιτική και να ε, αναλάβει και ε, να προσκαλέσει μάλλον και να έχει κάτω από την αιγίδα τη και την ε, Ευρωπαϊκή Εποπτεία Τραπεζών, τις οποίες τον επικεφαλή είχατε πριν από λίγο εδώ ενώπιον σα. Υπάρχει λοιπόν ο, η εποπτεία αυτή που είναι η νέα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας και ξέρουμε ότι έχουμε πετύχει βελτιώσεις, έχουν μειωθεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και οι περισσότερες ε, σημαντικές ε, τράπεζες έχουν μειώσει κατά το ίμιση τα μη ξεπεριτούμενα δάνεια που διαθέτουν. Όμως οι προκλήσεις παραμένουν και η Τραπεζική Ένωση και η Ένωση Κεφαλαιογορών πρέπει να ολοκληρωθούν και να υπάρχει έτσι βελτίωση όσον αφορά την πρόσβαση σε χρήμα. Υπάρχει χαμηλή κερδοφορία επίσης και το τοπίο αλλάζει συνεχώς γιατί οι μη τράπεζες απεκτούν όλο και σημαντικότερο ρόλο ως διαμεσολαβητές. Το μερίδιο των ε, μη τραπεζών σε σχέση με τις τράπεζες από 30% που ήταν πριν την κρίση σήμερα είναι 50%. Αυτές είναι τεράστιες αλλαγές που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όταν σκεφτόμαστε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι επιχειρήσεις δημοσιονομικής τεχνολογίας ε, επίσης έχουν το 1 τέταρτο του κλάδου στη διάθεσή του σήμερα. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον και οι κεντρικέ τράπεζε και οι επόπτε πρέπει να διασφαλίσουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά να είναι και ανοιχτοί σε ευκαιρίε που προσφέρουν οι αλλαγέ αυτέ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε γρήγορση όσον αφορά του ε, κινδύνου για να αποφεύγουμε ε, κλιματικές δραστηριότητες, να προστατεύουμε τον ιδιωτικό βίο, να διασφαλίζουμε την εφαρμογή των ε, ρυθμίσεων και να προστατεύουμε τα δημόσια αγαθά. Αλλά σημαίνει επίσης ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στα ωφέλη από τα οποία μπορεί να υποφεληθεί η κοινωνία εξαιτία καινοτομιών. Οπότε είπαμε δέσμευση, να είμαστε πιστοί στην εντολή μας, ε, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και κάτι άλλο που βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η συμμετοχή όλων, να μην υπάρχουν αποκλεισμοί και θα σα εξηγήσω τι ακριβώ εννοώ. Η πρώτη πτυχή του όρου αυτού κατά τη γνώμη μου είναι η συμμετοχή και η συνεργασία. Μέσα στο ευρωσύστημα υπάρχει πραγματογνωμοσύνη που μπορεί να μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε μελλοντικέ προκλήσεις. Ένα παράδειγμα είναι το πρασίνισμα των δημοσιονομικών. Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ε, για αυτό το σκοπό το 2017 που συμμετέχουν οι κεντρικοί τραπεζίτε και επόπτε και αποτελεί μέλο του δικτύου αυτού και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να γίνουν αλλαγέ. Οι κεντρικέ τράπεζε μπορούν επίση να παίξουν σημαντικό ρόλο προκειμένου να ενισχύσουν ε, την συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο και να βοηθήσουν την ε, πολυμερή τάξη σε όλου του τομεί των αρμοδιοτήτων οι κεντρικές τράπεζες δεν δρούν μέσα σε ένα κενό. Πρέπει να φροντίζουν για την ε, αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής, η οποία μπορεί να ενισχυθεί εφόσον έχουμε τις κατάλληλες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και εφόσον υπάρχει η εμπιστοσύνη του κοινού. Γι' αυτό λοιπόν βλέπω πολλά περιθώρια για παρετέρω συνεργασία σε πολλούς τομείς πολιτικής. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς επίσης, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, πρέπει να προχωρήσει, αλλά να διασφαλίσουμε επίσης και την προστασία των ε, καταναλωτών, αποφεύγοντας το κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτό ισχύει τόσο στην πραγματική οικονομία όσο και στι υπηρεσίε, αλλά και τον χρηματοπιστωτικό τομέα για τον οποίο μιλήσαμε πριν. Ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτη. Ένα άλλο τομέα συνεργασία είναι οι δημοσιονομικέ πολιτικέ, που πρέπει να βοηθούν τη σταθεροποίηση των οικονομιών μα και να αποφεύγουν τον υπερβολικό φόρτο στην νομισματική πολιτική. Όταν ήμουν Υπουργό Οικονομικών, διαπίστωσα τι δυσκολίε στο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών. Εμεί είμαστε επικεντρωμένοι στα εθνικά μα ζητήματα και ξεχνάμε τα άλλα. Όμως η ευρωπαϊκή διάσταση μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να ε, αποφεύγουμε τους τριγμούς εξαιτία εξωτερικών ε, σοκ. Και όλα αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία εγώ τα λέω έτσι από το κεφάλι μου. Έχω δουλέψει πάρα πολύ όσον αφορά την απλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των κανόνων που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση και την εμβάθυνση των αγορών. Βραχυπρόθεσμα, μετά τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και με την προστασία που έχουμε από το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και δημιουργώντας επίσης και άλλα δημοσιονομικά εργαλεία θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά. Σε συνδυασμό μάλιστα με άλλες μεταρρυθμίσεις στα συστήματα πληρωμών, αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν να ενισχύσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσει να υποφεληθεί ακόμα περισσότερο το ευρώ εφόσον αποτελέσει αποθεματικό σε διεθνές επίπεδο και θα μπορέσει να διατηρήσει περισσότερο την ανεξαρτησία του μέσα σε έναν όλο και περισσότερο βέβαιο κόσμο. Η δεύτερη διάσταση της ε, συμμετοχής, όπως έλεγα, είναι η ποικιλομορφία. Ο Πολ Βαλερή είχε πει ότι πρέπει να βάλουμε από κοινού ό,τι καλύτερο έχουμε και να πλουτίσουμε από τις διαφορές μας. Η Σιμών Βέιλ επίσης έκανε μια αντίστοιχη ε, παρατήρηση όταν ήταν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγώ πιστεύω ότι η ποικιλομορφία αποτελεί πλούτο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε ταλέντο, κάθε γνώση και πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως οφείλου, ε, φιλής, ε, υποβάθρου, προέλευσης και να ακούμε επίσης παντός είδους φωνές όσο γίνεται περισσότερο και να διασφαλίσουμε ότι ο διάλογος αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εκπόνησης πολιτικής. Και γι' αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ για το διάλογο που θα μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας εφόσον επιβεβαιωθώ επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να ακούει και πρέπει να καταλαβαίνει τις αγορές. Δεν πρέπει να την καθοδηγούν οι αγορές, όχι, αλλά να ακούει και να καταλαβαίνει Επίσης πρέπει να ακούει και να καταλαβαίνει τον κόσμο. Γιατί ένα νόμισμα αποτελεί ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο ανήκει στον κόσμο. Όταν ήμουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δούλεψα σκληρά προκειμένου οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών να συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δουλέψουμε σκληρά και να διασφαλίσουμε ότι οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και οι άνθρωποι ε, νιώθουν δικό τους το νόμισμα αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πιστεύω ότι μόνο αν έχουμε ένα ζωντανό διάλογο μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Συνεπώς, ε, πρέπει να έχουμε τη δέσμευση στις ε, Εντολέ τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρειάζεται προσαρμοστικότητα και χρειάζεται και συμμετοχή όλων. Χρειάζεται επικοινωνία. Προσβλέπω λοιπόν σε μια καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων μαζί σα και είμαι εδώ μόνο για να απαντήσω στις ερωτήσει σα. Έχω ετοιμαστεί σκληρά. Έχω την εμπειρία που έχω συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά είμαι εδώ για να ακούσω και τι δικέ σα τι απόψει. και για να καταλάβω τι εσεί περιμένετε από την επικεφαλή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σα ευχαριστώ πολύ. πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε, αλλά πρέπει να προσαρμόσουμε και το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Στον πρώτο γύρο ερωτήσεων, πέντε λεπτά για τον καθένα και μετά στον επόμενο γύρο ερωτήσεων θα δούμε πόσο χρόνο θα έχει ο καθένας. Ο κύριος Φέρμπερ, εκ μέρους του ΕΛΚ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα μου επιτρέψετε, ε, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω γερμανικά. Θα ήθελα εξ ονόματος του ΕΛΚ να σας καλωσορίσω θερμά, ε, ενδεχομένως σε μια νέα θέση ε, στην προηγούμενη θέση σας ε, είχατε έρθει επανειλημμένα, σας είχαμε δει εδώ, με γενικά λόγια μας παρουσιάσετε ποια είναι τα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και εγώ εκεί θέλω να εστιάσω στην εντολή που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη τελική ανάλυση. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που αποφασίζουν για άλλα θέματα, θέματα όμως που δεν έχουν καμία σχέση με τις αρμοδιότητες της ΕΚΤ. Εσείς λοιπόν είπατε ότι πρέπει κανείς να δει το πλωστάσιο των εργαλείων ε, που υπάρχουν την εργαλειοθήκη. Εγώ διάβασα μία μελέτη που προέκυψε κατά τη διάρκεια της σας και εκεί αναφέρεται ότι πρέπει να καταργηθούν οι συναλλαγές ε, μετρητά. Ε, θα πρέπει επίσης ε, να γίνεται σωστός υπολογισμός των υπολείπων. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα, ε, τι ακριβώς έχετε κατά νου όταν λέτε ότι θα πρέπει κανείς να εξετάσει και νέα καινοτόμα εργαλεία έτσι ώστε να υλοποιήσει την εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Uh, το 2008 και πιο συγκεκριμένα το 2014, πολύ λίγοι άνθρωποι θα περίμεναν να υπάρξουν κάποια εργαλεία ε, ορισμένα εξ αυτών ε, τα ανακάλυψε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είτε πρόκειτο για μακροπροληπτικά εργαλεία, είτε πρόκειτο για προγράμματα αγοράς ε, διαφόρων άλλων εργαλείων, είτε πρόκειτο για στοχευμένους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Νομίζω ότι ε, τότε κανείς δεν περίμενε ότι πολλοί θα ήταν αγκασμένοι να καταφύγουν σε άλλα εργαλεία. Έγινε λοιπόν πολλή δουλειά για να υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα της εποχής. Και προφανώς ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εστίασε στο να ανταποκριθεί στο 1.127 τη Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυρίως εστιάζει στην σταθερότητα των τιμών. Έχοντας λοιπόν κατά νου την σταθερότητα των τιμών χρησιμοποιήθηκε ένα οπλοστάσιο ε, έτσι ώστε να έχουμε ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ξέρετε είναι πάντα πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τις αντιδράσεις, γιατί σε όταν υπάρχουν συγκεκριμένε αντιδράσει, πρέπει κανείς πάντα να υπολογίζει τι θα γινόταν αν δεν είχαν χρησιμοποιηθεί αυτό το εργαλείο. Πάντως, εμείς προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε την αξία όλων αυτών των εργαλείων και είναι σαφές ε, ότι αυτά τα εργαλεία βοηθούν έτσι ώστε να αναπτυχθεί η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη το 2% είναι εκεί που έφτασε η ΕΚΤ και πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης προέκυψαν ως αποτέλεσμα αυτής της ανανεωμένης εμπιστοσύνης. Έχοντας το βλέμμα προς το μέλλον, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι απειλές, ποιες είναι οι συνθήκες, ε, ποια είναι τα πιο κατάλληλα εργαλεία από αυτά που έχουμε και μέσα στο περιθώριο που υπάρχει για να χρησιμοποιηθούν, ε, ποια είναι η ανάλυση κόστους-οφέλους στην χρήση αυτών των εργαλείων και μέχρι ποιο βαθμό. Πρόκειται λοιπόν σαφώς για αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται ε, συλλογικά από το ε, Προεδρείο μας, από το Διοικητικό μας Συμβούλιο. Δεν θέλω να πω τι θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου. Ε, δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ ενδεχομένω να συμμετέχω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να καθορίσω τίποτα. Εγώ Πιστεύω ότι η ανάλυση κόστους ωφέλους και ίσως και η αναθεώρηση ε, του νομισματικού πλαισίου που θα πρέπει να γίνει όχι μόνο από την ΕΚΤ αλλά και σε συνεργασία με, άλλους, με άλλες κεντρικές τράπεζες του κόσμου, αυτό είναι επιτιμητό λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν. Γιώνας Φερνάνδης, παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Η δική μου η ερώτηση που είχα προετοιμάσει μοιάζει πάρα πολύ με αυτή που έκανε ο κύριος Φέρμπερ, αλλά ίσως με κάποια διαφορετική απόκριση. Ε, στις γραπτές σας απαντήσεις σε αυτήν την Επιτροπή υπάρχει μία απάντηση που δίνεται και θέλω να διευκρινίσετε στην ερώτηση παριθμών 6 σχετικά με την δυνατότητα να προαχθούν ή όχι ε, τα νομισματικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς αναφέρεστε στις ε, αλλαγές ε, που έγιναν από την αρχή της κρίσης, αλλά δεν μας δίνεται μια ξεκάθαρη θετική ή αρνητική απάντηση. Το πλαίσιο υπάρχει από το 2003 πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση και χρησιμοποιήθηκε από την ΕΚΤ ως ένα συμπληρωματικό μέτρο. Έκτοτε όμως ε, μειώθηκαν τα επιτόκια και αυτό ε, προέκυψε στο να ε, μειωθούν και περιορισμοί από τις τράπεζες. Συμφωνώ με τον κύριο Φέρμπερ ότι πρέπει να αυξήσουμε το ε, πραγματικό, όχι το ονομαστικό επιτόκιο. Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση νομίζω ότι αξίζει να ε, δούμε λιγάκι το πλαίσιο, να το αναλύσουμε, να μελετήσουμε τα περιθώρια που υπάρχουν για την ε, αύξηση του ε, κανονικού, του κανονικού επιτοκίου και θα ήθελα να μας πείτε τι μπορεί να κάνει η ΕΚ σε περίπτωση πραγματικής κρίσης. Υπάρχουν οι στόχοι που έχουν αναφερθεί ή ενδεχομένως και η μελέτη κάποιας, ε, κάποιου ψηφιακού νομίσματος. Εσείς ε, στηρίζετε αυτό το νομισματικό πλαίσιο που έχει στηρίξει παραδείγματο χάρη η Τράπεζα του Καναδά ή η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών και μπορείτε να είστε λίγο πιο σαφείς από ό,τι στη γραπτή σας απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κοιτάξτε, στην γραπτή μου απάντηση προσπάθησα να είμαι ε, ουσιαστική να απαντήσω, αλλά θα επανέλθω στη δική σας την ερώτηση. Κοιτάξτε, από το 2003 έχει περάσει πάρα πολύ καιρός και από τότε έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά την ΕΚΤ. Αν δούμε λιγάκι άλλες κεντρικές τράπεζες που είναι αξιοσέβαστες με πολύ καλή φήμη, η Bank of Canada, η Τράπεζα του Καναδά, αλλάζει το ρυθμιστικό της πλαίσιο κάθε πέντε χρόνια. Η Fed των Πολιτειών ξεκίνησε μία αναθεώρηση του ε, ρυθμιστικού πλαισίου πριν από έξι μήνες και θα διαρκέσει 12 μήνες για να μπορέσει να λάβει υπόψη της όλους τους ενδιαφερόμενους να κάνει απολογισμό όλων των απόψεων που έχουν σχέση με το πλαίσιο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι με την ειν προεδρία του κυρίου Ντράγκη υπάρχουν ήδη κάποια στοιχεία επανεξέτασης κάποιων στοιχείων του νομισματικού πλαισίου. Έχω κατά νου κυρίως αυτά τα οποία ελέγχθησαν τον Ιούλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καθορίσουμε κατά πόσον ο πληθωρισμός που είναι κοντά ή κάτω από 2%, κατά πόσον ο πληθωρισμός θα πρέπει να επιτυγχάνεται από κάτω ή με ένα ασύμετρο τρόπο, κατά πόσον αυτός είναι ήδη ένας τρόπος για να ανεθωρηθούν στοιχεία του ε, νομισματικού πλαισίου. Πιστεύω λοιπόν ότι η διευκρίνηση του στόχου είναι κάτι ε, το οποίο έχει ήδη εξεταστεί. Ε, δεν είναι σαφές ακριβώς ποιος είναι ο στόχος. Σε τελική ανάλυση, ε, τι είναι κοντά στο 2%, μιλάμε 1,6 για 1,9. Υπάρχει ευελιξία και εγώ, εξ όσων μπορώ να καταλάβω αυτά που μας λέει ο πρόεδρος τουλάχιστον της ΕΚΤ, είναι ότι δεν είναι το 1,6. Δεν λέει ακριβώς τι είναι. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουν βρεθεί σε αρμοδιότητα κεντρικού τραπεζίτη καταλαβαίνουν πολύ καλά το πόσο λεπτό είναι όλο αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ήταν ο κεντρικός ε, τραπεζίτης ε, στην Αυστραλία, στο Jackson Hole, εκεί συναντήκαμε όλοι μας και εκείνος είπε ε, Καταλαβαίνει, πιστεύετε κανείς ένας μέσος άνθρωπος γιατί δαπανάμε τόσο πολύ χρόνο που να λέμε κοντά στο 2% αλλά όχι πάνω από τους 2%. Άρα δηλαδή πρώτον πρέπει να διευκρινίσουμε, να ερευνήσουμε, να συνυπολογίσουμε απόψεις, να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις και με βάση ανάλυση κόστους ωφέλους να διευκρινίσουμε καλύτερα το πλαίσιο. Εγώ ε, λοιπόν ενθαρρύνω και στηρίζω αυτήν την εξέλιξη εξέλιξη ε, και βεβαίως χρειάζεται η απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για να ληφθεί περαιτέρω απόφαση. Εκ μέρους του Renew Europe, ο κύριος Λουί Γκαρικάνο. Κύριε Λαγκάρντ, σα εύχομαι καλή επιτυχία με όλη την εμπειρία που έχετε και τι ικανότητε που έχετε για τη νέα θέση στην οποία έχετε οριστεί. Ζούμε σε δύσκολε εποχές. Ο λαϊκισμός και ο εμπορικός πόλεμος ε, που έχει ξεκινήσει από τον πρόεδρο Τραμπ και άλλα σοκ στην παγκόσμια οικονομία θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε νέα ύφεση. Αυτό που με απασχολεί και εμένα προσωπικά και πολλούς Ευρωπαίους πολίτες είναι ότι η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες. Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οι προκάτοχοί σας εξήγησαν ή σχεδόν εξήγησαν τα συμβατικά μέτρα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερο πεδίο για χαμηλότερα ή πολύ χαμηλότερα επιτόκια ή για ε, συνέχιση αυτής της νομισματικής πολιτικής. Πολλοί διερωτώνται αν υπάρχει περαιτέρω περιθώριο. Όσον αφορά την Ευρωζώνη, δεν έχουμε κάνει όλα όσα θα μπορούσαμε να κάνουμε. Έχουν γίνει πολλά διαρθρωτικά ε, ζητήματα πολλά δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει, δεν έχουμε ένα δημοσιονομικό εργαλείο για σταθεροποίηση της οικονομίας, πολλά δεν έχουν γίνει. Οι ερωτήσεις μου λοιπόν είναι δύο στους δύο αυτούς τομείς. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να καταπολεμήσει μια πιθανή νέα ύφεση. Σε αυτή την περίπτωση, τι εργαλεία χρησιμοποίησε στο παρελθόν, τι νέα εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Και δεύτερον, για την Ευρωζώνη έχει κάνει η Ευρωζώνη ότι μπορούσε να κάνει μέχρι τώρα. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες. Τι νομίζετε ότι θα έπρεπε να κάνει το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και πώς βλέπετε το δικό σας ρόλο στο να προωθήσετε αυτά τα οποία πρέπει να κάνει η Ευρωζώνη. Είτε πρόκειται για ασφάλιση καταθέσεων, είτε μηχανισμός ασφαλείας, διάσωσης. Ευχαριστώ. Κύριε Λαγκάντε, ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια στην αρχή. Θυμάμαι στην εποχή της κρίσης, πολλοί διοικητέ κεντρικών τραπεζών διαμαρτύρονταν λέγοντας ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να δώσει λύση. Και βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι διοικητές κεντρικών τραπεζών χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία που έχουν στην εργαλειοθήκη τους, ε, ε, χρησιμοποιούν και επανεξετάζουν όλες τις πολιτικές κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα διαθέσιμα εργαλεία και αυτό πρέπει να κάνουν σύμφωνα με την ε, εντολή που έχουν. Σαφώς ε, πρέπει να υπάρχει συνεργασία και όλα τα θεσμικά όργανα στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη συγκεκριμένα για να ανταποκριθούμε στις απειλές ε, του λαϊκισμού πρέπει να υπάρξει τέτοια συνεργασία. Ε, ε, όταν και αν γίνω πρόεδρος ε, της ΕΚΤ υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε για το ρόλο που μπορούν να παίξουν πολλές χώρες. Το έχω πει πολλές φορές ως επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι ορισμένες χώρες στην Ευρωζώνη μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημοσιονομικό χώρο που έχουν για να βελτιώσουν τις υποδομές, τις τα ευρυζωνικά δίκτυα, να καταπολεμήσουν δηλαδή ε, τις πηγές ύφεση. Και υπάρχουν όλο και περισσότερες χώρες σήμερα. Αν δείτε τις χώρες της Ευρωζώνης, αν δείτε τις χώρες που βρίσκονται περίπου σε μηδενικό έλλειμμα ή με 0,5% έλλειμμα, οι περισσότερες χώρες στην Ευρωζώνη είναι σε αυτή τη θέση. Άρα, σαφώς δεν υπάρχει μεγάλο πεδίο, αλλά υπάρχει πεδίο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις δημοσιονομικές πολιτικές. Δεύτερον, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε πάρα πολλές χώρες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σε μερικές χώρες έχουν ξεκινήσει, κάποιες μεταρρυθμίσεις ε, έχουν εξεταστεί χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα όμως και σαφώς οι χώρες που δεν έχουν το δημοσιονομικό χώρο σήμερα, λιγότερο από το ίμιση των χωρών της Ευρωζώνης, πρέπει να επανασχεδιάσουν ε, το μείγμα δημοσιονομικών πολιτικών και πολιτικών υπέρ της ανάπτυξης, ε, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, γιατί αυτές είναι οι συνθήκες στις οποίες μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές μεταρρυθμίσεις καλύτερα και να δώσουν καλύτερα αποτελέσματα τώρα που υπάρχει κάποια ανάπτυξη. Το σωστό μείγμα λοιπόν κατάλληλης νομισματικής πολιτικής με όλα τα διαθέσιμα μέσα, νομισματικές, ε, δημοσιονομικές συγγνώμη, πολιτικές με τις χώρες που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις παράλληλα. Σβέν Γκίγκολ, εκ των Πρασίνων. Σας ευχαριστώ. Κυρία Λαγκάρντ, καταρχήν θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την οποία είστε υποψήφια ε, να γίνεται πρόεδρος. Είναι μια, ένα, ένα θεσμικό όργανο ιδιαίτερα ισχυρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι καλό μήνυμα, καλό ιονό το ότι μια ισχυρή γυναίκα θέτει υποψηφιότητα για ένα ισχυρό οργανισμό και θα ήταν καλό αυτό ο ισχυρό οργανισμό ε, να έχει επικεφαλής μια γυναίκα. Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από άνδρες είναι καλό να έχουμε γυναίκε υποψηφίου για τέτοιε θέσει. Πέραν τούτου θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αυτή που έσωσε το ευρώ και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όχι πολιτικοί άνδρες και γυναίκες, αλλά η ΕΚΤ έσωσε το ευρώ. και μετά την νομισματική πολιτική επήλθε ένα επίπεδο λαϊκισμού πάρα πολύ υψηλό οι πολιτικοί δεν έκαναν τη δουλειά τους και χρειάστηκε από την ΕΚΤ παρέμβαση για στενότερη συνεργασία, για δημιουργία ενιαίας αγοράς και καλύτερη συνεργασία στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος που η ΕΚΤ έπρεπε να είναι επιθετική στην νομισματική της πολιτική. Και το είπατε κι εσείς ότι τα βλέπετε τα προβλήματα, βλέπετε τις ανησυχίες των πολιτών λόγω των αρνητικών παρενεργειών της επιθετικής πολιτικής είχα την εντύπωση ότι ο προκάτοχός σας δεν επικοινωνούσε με όλους τους πολίτες, δεν προσπαθούσε να εξηγήσει με πιστικό τρόπο γιατί απαιτούνται αυτά τα μέτρα που λαμβάνονταν. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις τις οποίες είδατε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους πολίτες και να εξηγήσετε τις αρνητικές επιπτώσεις. Αναφέρεται επίσης και το πρασίνισμα τη χρηματοπιστωτικής πολιτικής. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρχει χρηματοπιστωτική και νομισματική σταθερότητα χωρίς καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και η ΕΚΤ πρέπει να παίξει το ρόλο της γιατί είναι το πιο ισχυρό χρηματοπιστωτικό όργανο. Στις απαντήσεις σας λέτε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο μπορεί να το κάνει. Δεν είναι αρκετά ισχυρή η διατύπωση στην απάντησή σας. Μπορείτε να είστε πιο στεναροί και πιο τολμηροί σε αυτό το πρασίνισμα της χρηματοπιστωτικής πολιτικής υπό την ηγεσία σας στην ΕΚΤ απάντηση. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω την προσωπική μου θέση για το θέμα αυτό και το κάνω με προσοχή γιατί δεν θέλω με αυτά που λέω να δεσμεύσω το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γιατί εγώ απλώς ε, είμαι υποψήφια για τη θέση, δεν είμαι πρόεδρος της ΕΚΤ. Η προσωπική μου θέση για αυτά τα θέματα είναι ότι σε οποιοδήποτε θεσμικό όργανο οι κίνδυνοι για από την κλιματική αλλαγή ε, και για την προστασία του κλίματος πρέπει να βρίσκονται ως βασική προτεραιότητα. Βεβαίως σταθερότητα, αλλά θα πρέπει ε, και η κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι για το περιβάλλον να θεωρούνται βασική αποστολή όλων των θεσμικών οργάνων. Και πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το, το σπίτι του ο καθένας για να μπορέσει να προχωρήσει και πιο πέρα να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτό ίσχυε και όσο ήμουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και θα μιλήσω για το ΔΝΤΟΥ πριν μιλήσω και για την ΕΚΤ. Κλιματικός κίνδυνο λοιπόν, αλληλεγγύε για το περιβάλλον και το δημοσιονομικό τμήμα και πολλά άλλα τμήματα, πολλέ άλλες διευθύνσει του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επικέντρωσαν την προσοχή του σε ε, ενισχύσει που δίδονταν, παραδείγματο χάρη για τα ορυκτά καύσιμα, το άμεσο και το έμεσο κόστο αυτών των ενισχύσεων. Επικεντρωθήκαμε επίση ε, σε προπολογισμού που θα έπρεπε να είναι δημοσιονομικά υπεύθυνοι. Αυτά για το Διεθνές Ταμείο. Τώρα για την ΕΚΤ, χωρίς να προδικάζω τι μπορεί να συμβεί, γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τελικά υπό την ηγεσία ε, του ε, Προέδρου. Και πάλι, όπως και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έτσι και για την ΕΚΤ, πρέπει να ξεκινήσουμε από τον ίδιο μας ε, τον οργανισμό για να ληφθούν οι αποφάσει ε, για το πού θα επενδύσει ο κάθε οργανισμός και για το πρασίνισμα του δικτύου. Όταν υπάρχουν οι διοικητέ κεντρικών τραπεζών ε, που λένε ότι οι αλλαγές ε, στο κλίμα είναι βασική κίνδυνη που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες, αν το άκουγα αυτό ω τράπεζα θα ανησυχούσα και θα άρχιζα να κοιτάζω τι προβλέψει μου. Θα άρχιζα να επανεξετάζω το, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Όσον αφορά τις επενδύσεις, και δεν θα μακρηγορήσω, η ΕΚΤ δεν μπορεί αποκλειστικά και μόνο να επενδύει. 2,6 δισεκατομμύρια χαρτοφυλάκιο δεν μπορεί να επενδύει αποκλειστικά σε πράσινα ομόλογα, διότι δεν ε, υπάρχουν αρκετά ε, στην αγορά. Αλλά αν δώσει ε, μηνύματα ότι θα μπορέσει να επενδύσει και η αγορά θα το καταγράψει και επομένως οι κατευθύνσεις των επενδύσεων θα έχουν κάποια ένδειξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Έχω μία ερώτηση. Αναφερθήκατε λίγο στην αρχική σας παρουσίαση. Πολλά υπόθηκαν για τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε και έχουμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο επιθετικές αυτοκρατορίες την αμερικανική με το δολάριο και την ε, κινέζικη, που προσπαθούν να επιτεθούν και μία και άλλη. Λοιπόν, στις διεθνείς συναλλαγές, τι εργαλεία έχουμε οι κεντρικές τράπεζες. Δεν θα έπρεπε να είχαμε κάτι υπέρ της ανεξαρτησίας των χωρών μελών. Και στα πλαίσια της εντολής σας, πώς φαντάζεστε, τι φαντάζεστε ότι θα κάνετε προκειμένου το ευρώ να γίνει διεθνές νόμισμα, ε, για τις συναλλαγές ή ως ε, αποθεματικό όπως θα έπρεπε να είναι και πώς το τραπεζικό σύστημα ε, θα είναι αντοχής για να μπορεί να αποφύγει τις επιθέσεις αυτές των αυτοκρατοριών. Είχα και μια άλλη ερώτηση, την οποία βέβαια σε ένα μεγάλο μέρος απαντήσατε. Εγώ θεωρώ ότι η αξιοπιστή ενός νομισματικού συστήματος εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτό το σύστημα και στις ικανότητές του να ανταποκριθεί στις ε, προσδοκίες. Είναι ξεκάθαρο όμως και το είπατε και εσείς, η περιβαλλοντική κρίση τελικά και οι αντιπαραθέσεις στην ανθρωπότητα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Η αξιοπιστία πάντως του νομισματικού συστήματος με τι εργαλεία θα εξασφαλιστεί για να ξεπεράσουμε αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνη που έχει συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Η κυρία ευχαριστώ για την διτή αυτή ερώτηση. Για την πρώτη σας ερώτηση για το ευρώ. Ένα νόμισμα για νομισματικά αποθέματα και διεθνές νόμισμα να αναγνωριστεί έτσι και πώς θα κρατήσει τη θέση του ανάμεσα σε δύο αυτοκρατορίες που αντιπαρατήθενται αυτή την εποχή. Μα το ευρώ ήδη σήμερα είναι ένα νόμισμα στο οποίο υπάρχουν μεγάλα αποθέματα. Παρά τις όποιες προσπάθειες κάνουν άλλες κεντρικές τράπεζες ή άλλες αρχές, το δολάριο είναι το πρώτο, αλλά και αυτό αλλάζει. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πρέπει να προσφέρουμε στο ευρώ ε, τα μέσα που χρειάζεται ώστε να είναι πραγματικά ένα διεθνές νόμισμα και για πληρωμές αλλά και για καταθέσεις. Τα συστήματα πληρωμών πρέπει να είναι απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματικά. Επίσης, οι ευρωπαϊκές κεφαλαγορές επίσης θα πρέπει να είναι περισσότερο αναπτυγμένε από ό,τι είναι σήμερα. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον πρόεδρο Γκουαλτιέρη, γιατί ξέρω ότι έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στην ενίσχυση και στην ευάθυνση των κεφαλαγορών στην Ευρώπη αγορά κεφαλαίων που δεν είναι θέμα βέβαια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί βασικό στοιχείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Αν πολλαπλασιάσουμε τις πηγές χρηματοδότησης για όλους τους οικονομικούς φορείς και αν προσφέρουμε εναλλακτικέ στα τραπεζικά συστήματα, ενισχύουμε το ρόλο του ευρώ. Και υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να εξετάσουμε αλλά είναι πιο μακροπρόθεσμο, είναι να έχουμε στη διάθεσή μας ένα μέσο, γιατί έχουμε το Αμερικανικό θησαυροφυλάκιο που εξασφαλίζει αυτούς που ανησυχούν. Κάτι αντίστοιχο δεν έχουμε σήμερα στην Ευρώπη με αρκετό μέγεθος και αρκετό βάθος για την Ευρωζώνη που να είναι ε, να αντιστοιχεί στο μέγεθος της Ευρωζώνης. Τα μέσα πληρωμή είναι εξαιρετικά αυτά που διαθέτουμε, αλλά πρέπει να τα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο για τις κεφαλαγορές και για την ενίσχυση του οπλοστασίου που διαθέτουμε. Απλοποίηση, αποτελεσματικότητα ε, δημοσιονομικών πολιτικών που να είναι συντονισμένες μεταξύ τους, τραπεζική ένωση, ε, μηχανισμός ε, προστασίας καταθέσεων. Όλα αυτά θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το ρόλο του ευρώ ως ε, νόμισμα στο οποίο μαζεύονται καταθέσεις. Κάποιος Ρωμανός οικονομολόγος έλεγε ότι όλα αυτά γίνονται πολύ αργά μέχρι κάποια στιγμή που ξαφνικά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε τέτοιου είδους εξελίξεις. Ευχαριστούμε. Τώρα για το ECR, ο κύριος Σέπινγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω την ερώτησή μου στα Ολλανδικά, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να μάθω για τα αρνητικά επιτόκια. Είναι σαφές ε, ότι η κυρία Λαγκάρτ ακόμα δεν έχει οριστεί βέβαια επικεφαλής, οπότε αφήνει όλες τις εναλλακτικέ ανοιχτές. Όμως τι σημαίνει για τους αποταμιευτές, τους καταθέτες, τους συνταξιοδοτούμενους τα αρνητικά επιτόκια. Γιατί με αρνητικά επιτόκια καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όταν υπάρχει κάποιος πληθωρισμός και έπειτα πρέπει να δούμε και την κλιματική πολιτική. Οι αποταμιευτές είναι στριμωγμένοι στη γωνία, είναι θυμωμένοι, χάνουν. 3% σε 10 χρόνια έχουν χάσει το 1 τρίτο του κεφαλαίου τους που εξαφανίζεται, εξατμίζεται. Και αν αυτά όταν έχουμε μηδενικό επιτόκιο. Όταν αρχίσουμε με τα αρνητικά επιτόκια, τι θα γίνει. Ο κόσμος θα γυρίσει ανάποδα. Ξαφνικά θα γίνεται η βασίλισσα του ευρώ. Όμως φοβάμαι ότι με τα αρνητικά επιτόκια θα έχετε εναντίον σας ε, τους ε, ανθρώπους στο δρόμο. Οι αποταμιεύσεις πρέπει να επιβραβεύονται και όχι το αντίθετο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Δεν μιλάω Ολλανδικά, δυστυχώς, οπότε θα σας απαντήσω αγγλικά. Νομίζω ότι στην ερώτησή σας έχω δώσει δύο απαντήσεις νωρίτερα, απαντώντας άλλους. Πάντα πρέπει να κάνουμε την ανάλυση κόστους-οφέλους για να δούμε ποιο είναι το καλύτερο μέσο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τον ε, πολλαπλή ρόλο του πληθυσμού. Κάποιοι είναι δανειστές, κάποιοι δανείζουν, κάποιες χώρες μέλη είναι βαριά χρεωμένες, κάποιες άλλες όχι. Και οι επιπτώσεις του όποιου επιτοκίου εξαρτάται από το για ποιον μιλάμε. Όταν λοιπόν αναθεωρούμε το πλαίσιο και εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα των μέσων που έχουμε χρησιμοποιήσει, πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλους αυτούς τους ρόλους τις διαφορετικές περιπτώσεις και να αποφασίσουμε σε τι βαθμό και πόσο βαθιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια μέσα για να έχουν καθαρά θετικό αποτέλεσμα. Αν υπάρχει ύφεση, αν υπάρχει το αντίθετο, εξαρτάται από τον στόχο κάθε φορά και μην ξεχνάμε ότι αν διαπιστώσουμε ότι δεν είναι καλό για τον κόσμο, θα πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή. Πάντως, η νομισματική πολιτική με την προσφορά χρήματος είναι κάτι που χρειάζεται και θα χρειάζεται ακόμα για κάποιο καιρό. Και αυτό βέβαια χωρίς να ξέρουμε τι θα αποφασίσει τελικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα προς το παρόν. Και επιτρέψτε μου, γιατί έχω ένα λεπτό που θέλω να το χρησιμοποιήσω ακόμα. Πολύ σύντομα. Για αυτό που λέτε για τα θετικά και τα αρνητικά. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσω να βοηθήσω να κοινωνήσω το λόγο, το στόχο που προσπαθώ να πετύχω. Αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό θα προσπαθήσω να αναπτύξω όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Όχι αγορές, γιατί οι αγορές καταλαβαίνουν όλες τις γλώσσες, όλα τα αρχικά που συζητάμε και πετάμε δεξιά και αριστερά. Όχι. Ο κόσμος της Ευρωζώνης πρέπει να καταλάβει γιατί παίρνονται αποφάσεις που παίρνονται. Ποιο είναι το θετικό, ποιος είναι ο απότερος στόχος, ε, ποια θα είναι η ζημιά στην αρχή και το ωφέλει αργότερα. Σε αυτά τα πράγματα θέλω εγώ να σπαταλήσω ενέργεια και χρόνο. Τελευταία σε αυτόν τον πρώτο κύκλο. Κυρία Μανώ ε, Καλημέρα. Επανέρχομαι μετά την παρατηρήση του Σβέν. Όταν ε, ε, ομιλώ πρώτη γυναίκα ομιλήτρια, μπορώ κι εγώ να πω ότι είναι κρίμα που δεσπόζει η αντρική παρουσία σε τέτοιου τομεί. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για δύο βασικά θέματα την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η νομισματική πολιτική παίζει θεμελιώδη ρόλο για αυτά τα δύο θέματα. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Δούλευα μέχρι τώρα για μία μη κυβερνητική οργάνωση, την Oxfam, που είχε ως βασικό αντικείμενο την καταπολέμηση των ανισοτήτων και χρησιμοποιούσαμε ε, τις ε, δηλώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τα θέματα ανισοτήτων. Και πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντας το ερωτηματολόγιο απογοητεύτηκα κάπως γιατί βλέπω ότι η λέξη ανισότητα μόνο δύο φορές εμφανίζεται, ενώ η σταθερότητα των τιμών εμφανίζεται 28 φορές. Ε, ίσως ε, στις ε, απαντήσεις σας μας δίνετε και την εικόνα των προτεραιοτήτων σας. Πάνω από χίλια δις έχουν δοθεί στο ε, τραπεζικό σύστημα και ε, μόνο 230 ε, σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά. Τεράστια ποσά δόθηκαν σε τράπεζες, βοηθώντας την κερδοσκοπία στις χρηματαγορές. Και ο Μάριο Ντράγκη είπε ότι οι πλέον πλούσιοι επωφελούνται κατά πάσα από, από την ποσοτική χαλάρωση. Ε, τι συγκεκριμένα μέτρα είστε πρόθυμοι να πάρετε για να βελτιώσετε την πραγματική οικονομία ώστε να μην επιδεινωθούν οι ανισότητες. Ο στόχος του να περιοριστεί ο πληθωρισμός που δεν είναι πλέον προσαρμοσμένος στην οικονομική συγκυρία με χαμηλή ανάπτυξη και πληθωρισμό ε, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την ε, φούσκα της κερδοσκοπίας που είδαμε τα τελευταία χρόνια και πώς μπορούμε να ενσωματίσουμε και άλλες παραμέτρους και όχι μόνο τη σταθερότητα των, των τιμών. Ε, χαίρομαι για αυτά που διάβασα στο ερωτηματολόγιο, στις απαντήσεις που δώσατε. Μιλάτε για την πράσινη συμφωνία. Ε, και εδώ θέλω να κάνω δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι πώς μπορούμε να σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε τις μορφές ενέργειας που ρηπαίνουν γιατί ο ιδιωτικός δανεισμός έχει ωφελήσει κυρίως επιχειρήσεις που ρηπαίνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό και δεν λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια στη χρηματοδότηση της ΕΚΤ θα μας μιλήσετε για τα πράσινα ομόλογα, αλλά και εσείς θα αναγνωρίζετε ότι είναι περιορισμένο το μέγεθος της αγοράς και δεν πρέπει και να στρεβλώσουμε την αγορά. Επομένως, εδώ έχουμε και ένα παράδοξο. Και άλλο ένα ερώτημα, πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η οικολογική παρέμβαση, αυτή η μετάβαση προς μια πιο, ένα πιο οικολογικό μέλλον. 190 δις το χρόνο χρειάζονται για τη χρηματοδότηση. Μιλάτε για το ρόλο του δημοσίου τομέα και τη δημόσια χρηματοδότηση. Στη σελίδα 26 λέτε κάτι που μου με εξέπληξε, ότι τελικά η νομισματική πολιτική δεν είναι πανάκια, δεν είναι η βασική πολιτική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγή. Πώς μπορεί να αναπροσαρμοστεί η νομισματική πολιτική για την προοπτική τη κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Για την ερώτησή σας σχετικά με την καταπολέμηση των ανισοτήτων, όντως είναι ένας τομέας ε, στον οποίο αναλάβαμε δεσμεύσεις ε, στο Δουνουτού και δουλέψαμε πολύ με την Oxfam, ε, με φίλους με τους οποίους προσπαθήσαμε να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και για, τα δύο, και για τους δύο οργανισμούς, και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για την Oxfam. Είναι σαφές ότι η σταθερότητα των τιμών παραμένει η βασική έδρα της ΕΚΤ, το άρθρο 27 το λέει, το αναφέρει ως πρωταρχικό στόχο. Υπάρχει και δευτερεύον στόχος ε, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι απαραίτητα δευτερεύον γιατί μόλις έχουμε σταθερότητα των τιμών, μόλις το επιτύχουμε θα δούμε ποιοι είναι και ε, οι στόχοι των άλλων θεσμικών οργάνων ώστε να έχουμε κάποια εναρμόνιση. Ο στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί επομένως απολύτως να αποτελέσει στόχο και της ΕΚΤ στις πολιτικές της. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για την απάντησή μου σχετικά με το πρασίνισμα και το πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη. Τα πράσινα ομόλογα όντως είναι μικρά σε αριθμό και νομίζω ότι η ΕΚΤ ε, μέχρι τώρα έχει παίξει κάποιο ρόλο. Υπάρχει και ένα πολύ καλό ε, ε, έγγραφο επί του οποίου θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Πρέπει ε, να καθοριστεί τι αποτελεί πράσινη επένδυση και τι όχι. Μέχρι τώρα υπάρχει ταξινόμηση σε πολλά επίπεδα, αλλά χρειάζεται μια διευκρίνηση του τι ακριβώς ε, εννοούμε και η ΕΚΤ που κάνει δράσεις αναχρηματοδότησης ε, προϊόντων που φτάνουν σε περίοδο ρήμανσης θα δώσει τη δυνατότητα ε, να αλλάξει κατεύθυνση και να κατευθυνθεί προς πιο πράσινα προϊόντα. Θα συνεχίσω λοιπόν να εμβαθύνω σε αυτό το θέμα για να μπορούμε πώς η ΕΚΤ μπορεί να δράσει. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος ε, και για να υπάρχει ε, κάποιος βαθμός ε, ισότητας για όλους τους βουλευτές θα ήθελα να βάλουμε ένα όριο 4,5 λεπτών και παρακαλώ κάνετε σύντομες ερωτήσεις. Ο κύριος Ότμαρ Κάρας. Κυρία Λαγκάρτ, σας συγχαίρω για την, για πρόταση ορισμού. Για μένα ε, το θέμα της ECB, της ΕΚΤ, ε, δεν είναι κάτι που μας ανησυχεί, είναι κάτι που αποτελεί μέρος του προβλήματος. Εσείς ε, εξηγήσατε τις προκλήσεις που υπάρχουν. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, πώς προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε την παγκόσμια προοπτική σας. Η επιτυχία σας στη θέση της Προέδρου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και η συμμετοχή σας στους G20 και στα προγράμματα οικονομικής στήριξης σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, στην Τρόικα, όλα αυτά σας ενίσχυσαν και σας ενισχύουν στη θέση της υποψηφίου του ΕΚΤ. Κάποιοι πολιτικοί όλο και περισσότερο περισσότερο ε, λένε ότι η ΕΚΤ φταίει για πάρα πολλά δεινά, ε, η ΕΚΤ φταίει για την αποτυχία, επικρίνουν το χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων. Αυτή η κριτική ε, προσκρούει σε ότα ακόντων και θέλω να σας ρωτήσω πώς ακριβώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το έλλειμμα. Those are very broad questions. Thank you. Οι ερωτήσεις σας καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα. Ε, κοιτάξτε, το να γίνω πρόεδρος της ΕΚΤΑ, αυτό σημαίνει ότι θα φέρω μαζί μου και την εμπειρία που έχω συγκεντρώσει σε διάφορες θέσεις. Και αυτό που βίασα στους ε, G20, στις διάφορες αντίστοιχες των G7, όλα αυτά που διαπίστωσα είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα σε αυτές τις ομάδες, οποτεδήποτε εμφανίζονται και ακραίες προκλήσεις. Ε, βεβαίως δεν επιθυμώ να υπάρχουν τέτοιου είδους προκλήσεις, γιατί εγώ αναμφίβολα δεν επιθυμώ ε, να υπάρξει οικονομική κρίση απλά και μόνο για να δείξουμε ότι οι G20, οι G7 ε, κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εκείνο όμως ε, που θέλω είναι να συμβάλλω σε αυτό το αίσθημα του επίγοντος ε, παρότι αυτή τη στιγμή δεν πληττόμεθα από κρίση. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτό το αίσθημα του κατεπίγοντος θα συνεχίσει η αναβολή, η αναβλητικότητα και δεν το λέω αν θέλετε με τη μορφή κριτικής αλλά αυτό προκύπτει από τις πολιτικές εκλογές. Ε, οι άνθρωποι καταφεύγουν στο δικό τους το γνώριμο περιβάλλον, στα εθνικά τους συμφέροντα. Ε, περιορίζεται ο δημοσιονομικό του ή ο νομισματικός τους ορίζοντα και πιστεύουν ότι κάποιο άλλο θα βρεθεί για να κάνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ε, Έχοντα υπάρξει λοιπόν σε διάφορε θέσει ω υπουργό Οικονομικών, ω επικεφαλής του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου που προσπάθησα να εντοπίσω καλύτερη νομοθέτηση, καλύτερα μείγματα πολιτικής, ε, θέλω να πιστεύω ότι εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα καλύτερη συνεργασία να κατανοήσουμε καλύτερα της τις προτεραιότητες ε, των διαφόρων παικτών και ξέρετε δεν είμαι κάτι το εξοκοσμικό, όπως ίσως κάποιος υπενήχθηκε ε, προηγουμένως, αλλά και εγώ θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα είναι συλλογικά. Είτε μιλάμε για την κλιματική αλλαγή, για την χρηματοψηφιακή σταθερότητα, την κυβερνοαπειλή, ε, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, τη φορολογία, την ε, πολιτική ανταγωνισμό. Όλα αυτά πλέον είναι διεθνή γιατί η πραγματική οικονομία έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο της διεθνικότητας. Και για να ανταποκριθεί κανείς στο αίσθημα των πολιτών ότι η μοίρα τους δεν βρίσκεται πια στα χέρια τους και ότι οι εθνικοί ταγοί δεν μπορούν και αυτοί να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, για να το αποφύγουμε αυτό πρέπει να δώσουμε απαντήσει. Και νομίζω ότι το κοινό Κοινοβούλιο ε, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι. Ο κύριος Μαρκές από τους σοσιαλδημοκράτες. Καλημέρα σας κυρία Λαγκάρτ. Η νομισματική πολιτική αποδείχθηκε ότι είναι καθοριστική σημασία για τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης, ε, το 2012 ε, είπε ο κύριος Ντράγκη ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των, ε, του δημόσιου χρέους. Αυτό αφορούσε και μια χώρα σαν τη δική μου, την Πορτογαλία. Εσείς θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά εκλεγείτε πρόεδρος της ΕΚΤΕ και εσείς ε, θα παραμείνετε σε αυτό το δόγμα ότι θα κάνω ό,τι πρέπει πάση θυσία για να διαφυλάξω το ευρώ. Ίσως να χρειαστεί να εφαρμοστούν και αντισυμβατικές πολιτικές για να διαφυλαχθεί το ευρώ και ε, θεωρώ ότι πρέπει ε, για να επιτύχουμε το στόχο μας να ολοκληρώσουμε και το θεσμικό πλαίσιο. Το λέτε αυτό στις απαντήσεις σας. Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο, η Τραπεζική Ένωση, ε, κυρίως το ΕΝΤΙΣ, Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα της Ασφάλισης των Καταθέσεων, το ΕΝΤΙΣ. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω όσον αφορά την τα δημοσιονομικά στην Ευρωζώνη. Ε, τι ακριβώς ε, μέτρα προτίθεστε να λάβετε και αυτό που είναι πιο κρίσιμο για τη σταθεροποίηση, θέλω να ρωτήσω, εσείς πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να στηρίξετε ένα εργαλείο όπως ε, αυτό που στηρίζει ο προ, η πρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, δηλαδή ένα σύστημα για την ε, χορήγηση επιδομάτων, ανεργίας. Εσείς συμφωνείτε σε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ τον προτέρων για την απάντησή σας. Ναι, ο πρόεδρος θα μου πει ότι εσείς το φάγατε το χρόνο και εγώ δεν έχω χρόνο να απαντήσω. Όταν ο πρόεδρος Ντράγκη είπε ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να σώσουμε το ευρώ και πιστέψτε με αυτά που θα κάνουμε αρκούν, ήμουνα παρούσα. Ελπίζω να μην, να μου συμβεί εμένα, αλλά αν μου συμβεί θα το κάνω κι εγώ. Γιατί πιστεύω ότι οι υπόλοιποι δεν κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Επιπλέον θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όταν είπε ότι ό,τι και να χρειαστεί θα το κάνουμε, τελικά αυτό που σχεδιάστηκε ήταν το OMT που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Αυτό που προέκυψε είναι η σταθεροποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού ε, να μην είναι δυνατόν να παραλύει ο μηχανισμός ε, μέσα από άλλες εξωτερικές επιδράσεις, γιατί εγώ έχω κάνει την εμπειρία ότι όταν φτιάξαμε την, ε, όταν προέκυψε η κρίση να αντιμετωπίσαμε με, τα, με τους διάφορους θεσμούς που φτιάξαμε, ε, τότε δεν ανταποκριθήκαμε αρκετά γρήγορα. Αλλά αν τελικά εκλεγώ, εγώ θα προσπαθήσω να ασχοληθώ κυρίως με την σταθερότητα των τιμών. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά παρακλάδια, πολλές ε, προεκτάσεις ε, για να έχουμε μια σωστή πολιτική. Ως εκ τούτου θεωρώ και να σας πω ε, σχετικά με τις δημοσιονομικές μας αρμοδιότητες. Εμείς από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό που αναγνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα σε κάποια κράτη-μέλη, μεταξύ τους τα κράτη-μέλη. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά τι ακριβώς εννοώ. Και η δική μας η πρόταση είναι ότι μπορεί κανείς να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να υποβάλει αυστηρά stress test, να δεχτεί ένα εντονότερο βαθμό εποπτείας και έτσι λοιπόν το σύστημα εξασφάλισης καταθέσεων να ισχύει στο σύνολο της ε, Ευρωζώνης χωρίς κανένα περιορισμό. Το ίδιο ισχύει και για τη δημοσιονομική ικανότητα. Ε, εάν πρέπει να προχωρήσει περισσότερο και εκεί θα πρέπει να υφίστανται οι προϋποθέσεις που θα εγγυώνται ότι αν κάποιος καταθέσει τα χρήματά του σε μία χή χώρα, η χώρα αυτή ε, θα μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα σοκ, βεβαίως στο βαθμό που αυτή, αυτό το σοκ δεν είναι ενδυμικό. Ο κύριος Πασκάλ Καλφά. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ρωτήσω για την σχέση των δικών σας αρμοδιοτήτων και την κλιματική αλλαγή. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς αναφερθήκατε στις αναλύσεις του Μπένου Ακερέλ, που είναι τώρα κεντρικός τραπεζίτης, και είναι ήδη στην εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, το θέμα με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα σταθερότητα τιμών. Αν υπάρξει αλλαγή στο κλίμα 3-5 βαθμοί, σίγουρα θα υπάρξει αλλαγή και στις τιμές. Και επίσης είναι και το θέμα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ο Μακερνή και άλλοι τα έχουν πει ότι σήμερα δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μεσοπρόθεσμα χρηματοπιστωτική σταθερότητα αν δεν λάβουμε υπόψη μας το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Οι δύο ερωτήσεις μου. Πρώτον, δεσμεύεστε να χρησιμοποιήσετε την ταξινόμηση των επενδύσεων και του ενεργητικού σε πράσινα και μη πράσινα και να το λάβετε υπόψη σα. Δεύτερον, αναφερθήκατε στον απολογισμό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, όσον αφορά ε, τα πράσινα ομόλογα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, το κάθε ενεργειό και κάθε αγορά που έχει γίνει έχει να κάνει με τον άνθρακα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για πράσινε επενδύσει. Οπότε εσεί μπορείτε να μα πείτε ότι σιγά σιγά η ΕΚΤΕ θα αποδεσμευτεί από αυτό το ενεργητικό το οποίο είναι στεδεμένο άμεσα με τον άνθρακα. Και τρίτον, θα λάβετε υπόψη σας περισσότερο στις ε, μακροαναλύσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το θέμα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Απάντηση. Πρώτα απ' όλα, ελπίζω η ταξινόμηση των επενδύσεων που συζητάτε σήμερα θα καταλήξει σύντομα γιατί πιστεύω πραγματικά ότι είναι ένα βασικό στοιχείο που σήμερα αποτελεί τροχοπέδι σε διάφορα θέματα, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχω συμμετάσχει σε διάφορα φόρουμ, συζητήσει και με τον ιδιωτικό τομέα και με μεγάλου επενδυτέ. Βρίσκονται σε αβεβαιότητα όσον αφορά την ταξινόμηση αυτή την ιεράρχηση των προϊόντων σε πράσινα και λιγότερο πράσινα. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν ολοκληρωθεί η ταξινόμηση αυτή, τόσο το καλύτερο και όπω ε, και εσεί, όταν για πρώτη φορά φτάνετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι και εγώ είμαι αρχάρια για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, χρησιμοποιεί, θα χρησιμοποιήσει την ταξινόμηση αυτή στο μέλλον. Έτσι εκ προημίου δεν βλέπω γιατί να μην τηρήσει αυτό τον κανόνα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μου φαίνεται προφανές. Τώρα η σημερινοί βέβαια παράγοντες και φορείς θα μου πούν «Α, όχι, ουδετερότητα». Ναι, αλλά αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει μια τέτοια ταξινόμηση, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την ουδετερότητα. Θα υπερισχύει η ταξινόμηση δική σας στην ουδετερότητα. Τώρα για το μέγεθος του ενεργητικού των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τον άνθρακα. Ε, δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη, εννοείται. Αλλά το να πάμε σταδιακά ώστε να απαλείψουμε αυτού του είδου το ενεργητικό όπω συνδέεται με τον άνθρακα, ε, πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Είμαι πεπισμένη. Αν είμαστε πεπισμένοι για την απόλυτη αναγκαιότητα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποιο δεσμικό όργανο και αν βρισκόμαστε για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, πρέπει να το κάνουμε. Και προσθέτω και κάτι ακόμα. Στην ανάλυση κινδύνου που κάνουν οι κεντρικές τράπεζες πρέπει στην εποπτική τους αρμοδιότητα να λάβουν υπόψη τους και την κλιματική διάσταση, την προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι αποτελεί ένα μοχλό που δεν πρέπει να παραβλέψουμε όταν μιλάμε για προμήθειες, όταν μιλάμε για την εκτίμηση κινδύνου, οι τράπεζες πρέπει να το λάβουν υπόψη τους όταν προσδιορίζουν το κεφάλαιό τους. Ευχαριστούμε. Επόμενος ο μιλητής Διαφερέιρα από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λαγκάρτ, είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μια γυναίκα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είναι η πρώτη φορά που η εντολή της ε, Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ξεκινούν συγχρόνως. Είναι καλό. Όταν θα έχετε εκλεγεί θα μπορέσετε να συνεργαστείτε μεταξύ σας για να προχωρήσει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση που αυτό ακριβώ χρειαζόμαστε. Τώρα, στην τελευταία τη συνεδρία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούλιο αναφέρθηκαν μέτρα για την τόνωση τη ευρωπαϊκή οικονομία. Και κάποια μέλη τότε μίλησαν ενδεχομένω για ένα πακέτο μέτρο, όπως μείωση επιτοκίων και αγορά ενεργητικού. Τον Μάρτιο στην Πορτογαλία είπατε ότι πρέπει να αυξήσουμε την προσπάθεια για την μείωση του χρέους, ότι πρέπει δηλαδή να επισκευάζουμε τη σκεπή μας όταν έχουμε καλό καιρό και όχι όταν έχουμε κακό καιρό. Τώρα υπάρχουν χώρες με υψηλό χρέος όπως είναι η Πορτογαλία που εποφελήθηκαν από καλούς όρους για την χρηματοδότηση, επαναχρηματοδότηση του χρέους. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν από τον καλό καιρό εντό αγωγικών. Δεύτερον, η τεχνολογία, blockchain ή τα κρυπτονομίσματα, ε, παντός είδους τρόποι ε, πληρωμών Όλα αυτά υπάρχουν. Κάποιος από, το, από την Εκτελεστική Επιτροπή αναφέρθηκε στο Libra, ένα κρυπτονόμισμα ε, που κάποιες εταιρείες σκέφτονται να βάλουν στην αγορά και είπε ότι θα είναι απειλή αυτό. Ποια είναι η καλή ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα του συστήματος και σε κίνητρα για καινοτομία στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Απάντηση. Ευχαριστώ. Ναι, να επισκευάζουμε τη σκεπή όταν ε, ο καιρός είναι καλός. Ο Φιτζελ Κέναντι το είχε πει. Όντως, πολλοί χρησιμοποίησαν αυτή τη φράση, πολύ πολιτικοί και άλλοι. Αλλά πολλοί μείναν στα λόγια και δεν το έκαναν πράξη. Όσο υπάρχει ακόμα ανάπτυξη τώρα, και έχουμε περάσει από μια τεράστια περίοδο ανάπτυξης χωρίς προηγούμενο ε, σε πάρα πολλές χώρες. Και μετά έχουμε απειλές, είτε πρόκειται για το διεθνές εμπόριο, είτε υπάρχει το Brexit, είναι γεωπολιτική κίνδυνη. Για να μην αναφερθώ και στο κλίμα, τα είπαμε αυτά, που είναι πιο μακροχρόνιο θέμα, αλλά απαιτεί άμεσες λύσεις, ε, όντως ισχύει αυτό, το ότι πρέπει να επισκευάζουμε τη σκεπή του σπιτιού μας όταν ο καιρό είναι ακόμα καλός. Άλλες χώρες έχουν μεγάλα περιθώρια, άλλες πρέπει να προσαρμόσουν την πολιτική τους και να διευκολύνουν τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται. Τώρα για το δεύτερο ερώτημά σας που απαιτεί συζήτηση σε βάθος το θέμα των τεχνολογικών αλλαγών και ισορροπία ανάμεσα στο κόστος και στο όφελος από τέτοιες τεχνολογικές αλλαγές. Η γενική αρχή είναι ότι οι κυβερνήτες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να γνωρίζουν τις εξελίξεις, να ενημερώνονται συνεχώς, γιατί οι αλλαγές λαμβάνουν χώρα καθημερινά και πρέπει να το κάνουν αυτό έχοντας υπόψη στα εξή δύο. Πρώτον, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και προστασία καταναλωτών και επενδυτών. Και δεύτερον, να έχουν υπόψη τους να διευκολύνουν και να επιτρέπουν την καινοτομία. Γιατί οι κεντρικοί τραπεζίτες, όπως και άλλοι πολιτικοί, δεν μπορεί να κλείνουν τα μάτια και να παριστάνουν σαν να πρόκειται να συνεχιστούν τα πράγματα χωρίς καμία αλλαγή δεν είναι δυνατόν ε, να πηγαίνουν ε, με τον ίδιο τρόπο και να ταξιδεύουν ε, παντού νομίζοντας ότι θα συναντήσουν παντού τις ίδιες συνθήκες. Όχι, η τεχνολογία προχωράει, οι αλλαγές γίνονται. Και το ίδιο ισχύει και για την έκτη. Ποια από σας ξέρετε τα tips. Ακριβώς αυτό φοβόμουν. Ούτε εγώ ήξερα τι είναι τα tips. Είναι ένα σύστημα που το Νοέμβριο εγκαθίδρυσε η ΕΚΤ που δεν έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία ακόμα, όμως έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει απευθείας πληρωμές σε πραγματικό χρόνο μεταξύ ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό, θα δούμε αν οι τράπεζες θα το χρησιμοποιήσουν, αλλά είπαμε χρηματοπιστωτική σταθερότητα και καινοτομία. Και να θέτουμε το ερώτημα, πρέπει οι κεντρικές τράπεζες να είναι εκείνες που βρίσκονται στην αρχή τέτοιων τεχνολογικών επιτεγμάτων όπως τα κρυπτονομίσματα. Πολ Τάγκ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επανέλθω στο θέμα της δημοσιονομικής ικανότητας. Με ενδιαφέρει γιατί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, ήθελε να υπάρχει μια τέτοια, να υπάρχει δημοσιονομική ικανότητα και θέσατε και συγκεκριμένου όρου. Θεωρείτε ότι η καθυστέρηση τη εισαγωγή δημοσιονομική ικανότητα μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τη μακροοικονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη πέραν των όρων και προποθέσεων που θέσατε. Κάνω αυτή την πολύ συγκεκριμένη ερώτηση σε εσά. Το χρειαζόμαστε ή υπάρχουν κίνδυνοι για την μακροοικονομική σταθερότητα. Ε, δεύτερον, ε, για την Ελλάδα, ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι ο στόχος για το, ε, πλεόνασμα, για το πλεόνασμα είναι μη ρεαλιστικός και μη βιώσιμος και, και το θέμα της ελάφρυνση του χρέους. Συνεχίζετε να πιστεύετε αυτά τα οποία έχει πει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αν ναι, ως πρόεδρος της ΕΚΤ, Πώ θα τα χειριστείτε. Τρίτον, χαιρετίζω την έμφαση που θέσατε στη βιωσιμότητα. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και η ΕΚΤ ε, είναι ένα υπόδειγμα και έχει ένα ρόλο να παίξει για την βιώσιμη χρηματοδότηση. Η ΕΚΤ μπορεί να χρησιμοποιήσει το γενικό στόχο σύμφωνα με το άρθρο 127 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα ε, για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και το κλίμα. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ο πρωταρχικός στόχος αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει ε, θέσει σε προτεραιότητα τους δευτερογενείς στόχους για την καταπολέμηση του κλίματος. Εσείς θα υποστηρίξετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Απαντώντα πολύ άμεσα, δεν νομίζω ότι αν δεν ε, υλοποιήσουμε αυτόν ε, το μηχανισμό σταθερότητας που εγκρίθηκε αλλά δεν έχει προσδιοριστεί και δεν ε, έχουν οριστεί και συγκεκριμένα ποσά από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών τον Ιούνιο, δεν πρόκειται να κάνει να καταρρεύσει η σταθερότητα της Ευρωζώνης. Παρομοίως, Πιστεύω ότι για να ενδυναμωθεί και για να μπορέσει να αποτελέσει πραγματικά νομισματική ζώνη με όλα τα γνωρίσματα μιας νομισματικής ζώνης, θα είναι πολύ χρήσιμο και επιθυμητό να έχουμε αυτή τη δημοσιονομική σταθερότητα, όχι μόνο για λόγους ε, ε, σύγκλησης που είναι επιθυμητό στόχος, αλλά διότι ε, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα σοκ και τα προβλήματα, προβλήματα ρευστότητας. η μακροσταθερότητα θα επιβιώσει ακόμη και αν δεν το έχουμε τώρα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το χρειαστούμε στο μέλλον. Για την Ελλάδα και το πρωτογενέ πλεόνασμα είναι μια συζήτηση που συνεχίστηκε με την Τρόικα επί πολύ, ιδίω τα τελευταία χρόνια τη συμμετοχή του Δουνουτού στο πρόγραμμα. Και νομίζω ότι συνεχώ το Δουνουτού έλεγε ότι το 3,5% πρωτογενέ πλεόνασμα, κατά τη γνώμη του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και ακόμη μιλώ ω Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, είναι υπερβολικό στόχο και θέτει υπερβολική πίεση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, την οποία ελπίζαμε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συνεχίζει να έχει την άποψη αυτή και βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι σε περίοδο ανάκαμψης ε, και ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επανεξετάσουμε με μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι η δική μου αξιολόγηση. Ε, είναι πολύ χρήσιμο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρησε ε, το ρόλο της ΕΚΤ σε σχέση με τα προγράμματα, γιατί θυμάμαι ε, τις τεράστιες αυτές συναντήσεις, ατελείωτες συναντήσεις της Ευρωζώνης με άπειρες λεπτομέρειες για το είδος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ο Μάριο Ντράγκη και ε, οι υπάλληλοι της ΕΚΤ που ήταν ε, ε, στην αίθουσα συμμετείχαν. Και πραγματικά τίθεται το ερώτημα τι μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν ήταν η βασική τους αρμοδιότητα. Στο μέλλον η ΕΚΤ θα, θα περιορίζει την εξέτασή της στους τομείς που έχει αρμοδιότητα. Δεν έχουμε πλέον χρόνο, λέει ο Πρόεδρος. Ίσως ε, αργότερα μπορείτε να επανέλθετε. Νταμιάν καρέ εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ, κυρία Λαγκάρντ. Περιμένοντας λοιπόν ε, ε, να εφαρμοστεί αυτή η ευρωπαϊκή ταξινομία που αναφέρατε και με βάση και ε, τις κλιματικές εξελίξεις είστε πρόθυμοι να δεσμευτείτε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δημιουργήσετε μια πράσινη μεθοδολογία στο ΕΚΤ για το πρόγραμμα ενεργητικών λαμβάνοντας υπόψη και τις επιχειρήσεις που ρηπαίνουν περισσότερο και αποσύροντας σιγά σιγά τις επενδύσεις ε, της ΕΚΤ ε, από τις ε, επιχειρήσεις που ρηπαίνουν. Το 63% των χρηματοδοτήσεων πηγαίνουν σε επιχειρήσεις οι οποίες ρηπαίνουν, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες. Η ΕΚΤ έχει τακτικές συναντήσεις με τους επικεφαλής των μεγάλων τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά δεν έχει μια πλατφόρμα διαρθρωμένου διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών θα δεχόσατε να δημιουργηθεί ένα ετήσιο φόρουμ συζητήσεων στο πλαίσιο του οποίου η ΕΚΤ και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα μπορούσαν να συζητούν την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ως εκπρόσωπος της, όπως μας ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι της Φινλανδική Προεδρίας, ε, δεσμεύεστε να αναθεωρήσετε τους ε, κανόνες ηθικής και διοντολογία της ΕΚΤ για την ε, δημοσιοποίηση των συναντήσεων τη ΕΚΤ με λόμπι και με όλους τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών που σήμερα δεν δημοσιοποιούνται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την τελευταία σας ερώτηση, ξέρω ότι ο κώδικας δεοντολογίας αναθεωρήθηκε εις βάθος μετά από κάποια σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με τους εκπροσώπους ιδιωτικού τομέα. Χαίρομαι που ισχύουν οι σωστοί κανόνες του κώδικα διοντολογίας και θα ήθελα να εφαρμόζονται στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς εφαρμόζονται στην ιεραρχία της ΕΚΤ. Όσο καλύτερα και ε, με όσο μεγαλύτερη διαφάνεια εφαρμόζονται, τόσο καλύτερα για την τήρηση των αρχών της διοντολογίας για να διευκολύνεται και το είδος των επαφών και η ημερήσια διάταξη αυτών των συναντήσεων. Δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή καμία συγκεκριμένη δέσμευση, γιατί ε, ακόμη δεν ε, είμαι επικεφαλής της ΕΚΤ. Τώρα, για ένα ετήσιο φόρουμ. Και πάλι δεν μπορώ να δώσω δεσμεύσεις πρόορες, γιατί δεν βρίσκομαι ακόμη στη θέση της επικεφαλής της ΕΚΤ. Ε, όταν ήμουν στο Δουνουτού, αυτό το οποίο υλοποιήσαμε ε, ήταν ε, πολύ εντατικέ διαβουλεύσει τέτοιου τύπου. Και όσοι γνωρίζουν τι εργασίε του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου ξέρουν ότι πριν από 10 χρόνια οι εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών ήταν έξω από το Ταμείο και δημιουργήθηκε ένας επικοδομητικός διάλογος και δεν συμφωνούσαμε ούτε συμφωνούμε πάντοτε απολύτως. Αλλά καταφέραμε μέσω αυτού του επικοδομητικού διαλόγου να βρούμε ε, ε, τρόπο συνεννόησης ε, με τους εκπροσώπους τη κοινωνία των πολιτών από 189 χώρες ολόκληρου του κόσμου. Στην ετήσια συνέλευση του Δουνουτού, επί τρει ημέρες γίνεται αυτός ο διάλογος με κατανάλωση ενέργειας και με μεγάλο ενθουσιασμό. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η ανταλλαγή εμπειριών και ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών ήταν θεμελιώδους σημασία για να κατανοήσουμε καλύτερα τις προσδοκίες της ε, κοινωνίας των πολιτών, για να εξηγήσουμε καλύτερα τι είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, ποια είναι τα όρια των δράσεών μας και για να μπορέσουμε ε, να προωθήσουμε τις δράσεις μας χάρη στους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Όσον αφορά τη μεθοδολογία, Εάν ε, εφαρμόζεται μια ταξινομία η οποία εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να δούμε τη διαδικασία της ε, υλοποίησης αυτής της ταξινομίας και το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το ισοζύγιο ε, εκπομπών άνθρακα και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις επενδύσεις για εταιρείε όταν φτάνουν σε περίοδο ορίμανσης οι επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Γκούνερ Μπέκ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, ε, πιστεύω να ε, οριστείτε στην θέση της ε, Προέδρου της ε, ΕΚΤ. Σας καλωσορίζουμε καταρχήν εδώ. Θέλω να πω το εξή. Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν την, τον αναλάβουν όλοι από κοινού δημόσιο χρέος και απαγορεύουν και τη χρηματοδότηση από το κράτος είτε μέσα από εξαγορά ομολόγων είτε μέσα από άλλες κινήσεις απαγορεύεται και η αγορά δευτερογενών ε, ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Παρ' όλα αυτά, από το 2010 και κυρίως ε, από τότε που ε, ανέλαβε ο ακόμα πρόεδρος της ΕΚ, ο κύριος Ντράγκη, παρ' όλα αυτά, αυτά γίνονται. Ως Γαλλίδα Υπουργό ε, το 2010 και το 2011 είπατε τότε με δική σας πρωτοβουλία και πραγματικά τότε εγώ το είχα εκτιμήσει ιδιαίτερα και το εκτιμώ ακόμα. Είχατε πει λοιπόν ότι κατά την άποψή σας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και η ΕΚΤ έσπασαν, παραβίασαν τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, σώσουν το ευρώ και δεν είσαστε μόνο μία πολύ επιτυχημένη πολιτικός, αλλά και μία ε, νομικός εγνωσμένου κύρους. Γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, αν ε, συνεχίσετε, όπως και η προκάτοχή σας, να παραβιάζετε το δίκαιο, παραδείγματο χάρη ε, παρά τη συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευκολύνετε και να προβλέπετε ελαφρύνσεις για κράτη και επιχειρήσεις, τότε η σταθερότητα των τιμών κάτι για το οποίο έχετε δεσμευτεί, όπως επίσης και το 2% πληθωρισμός, κατά προσέγγιση 2%, ε, θα μπορούσε, όπως είπατε σήμερα, να ξεπεράσει και το 2%. Ε, κατ' ουσίαν, Όλα αυτά τι σημαίνουν. Σημαίνουν ότι οι καταθέτες, οι φορολογούμενοι και πολλοί άλλοι, οι οποίοι φέρουν τη λιγότερη ευθύνη για την κρίση, αυτοί θα επιβαρυνθούν. Και ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η αρχή της ίδιας ευθύνης στα δημοσιονομικά που και αυτή υπονομεύεται. Και ένα άλλο ερώτημα. Σε τελική ανάλυση, εσείς πώς αιτιολογείτε το δικαίωμα το οποίο διεκδίκησε η ΕΚΤ να είναι πάνω από οποιοδήποτε μορφή δικαίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί ε, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο και υπάρχουν πολλοί αρμόδιοι οι οποίοι προσπαθούν να εντοπίσουν το τι είναι νόμιμο και τι καθίσταται παράνομο. Νομίζω μέσα ακριβώς αυτά τα όρια πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν οι θεσμοί. Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά αρκετές φορές και σε διεθνές και σε περιφερειακό επίπεδο αναγκαστήκαμε να αποκλίνουμε, δεν θα έλεγα απαραίτητα να παραβιάσουμε τις συνθήκες, γιατί υπήρχαν ε, τομείς και θέματα όπου δεν υπήρχαν προβλέψεις, δεν είχε τίποτα προβλεφτεί το τι πρέπει να γίνει για να ε, προστατευτούν παραδείγματος χάρη οι καταθέσεις και οι αποταμιεύσεις των καταθετών. Το 8-9 σχεδόν όλοι είχαν προχωρήσει πέρα από τους κανόνες και αυτό για το κοινό καλό. Γιατί, για να μην χάσουν οι άνθρωποι τις καταθέσεις τους. Ακούω πολύ συχνά αυτούς που μας λένε ότι προστατεύσατε το χρηματοψηφιακό σύστημα. Όχι, δεν είναι έτσι. Εμείς απλά διασφαλίσαμε να μην υπάρξει πανικός, τραπεζικός πανικός, ε, να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες για να προστατευτούν οι καταθέσεις. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και δικαιολογημένο και απαραίτητο. Όσον αφορά τώρα το 2%, ε, κάτω από αλλά κοντά στο 2%, αυτό που συζητιέται στην ΕΚΤ ε, είναι το εξής. Μπορεί να πλησιάσει κανείς το 2% από κάτω, ανεβαίνοντα σιγά σιγά, 1,678, αλλά μπορεί να πάει στο 2% και από πάνω. Και νομίζω ότι αυτό το μεσοσταθμικό το 2% έτσι πρέπει να το ερμηνεύεται. Τουλάχιστον εγώ έτσι κατανοώ και ερμηνεύω τη συζήτηση και είναι σωστό να υπάρχει μια συμφωνία που είναι αποδεκτή και από επάνω αλλά και από κάτω. Επόμενος ομιλητής από το ECR. Χαίρομαι που σας βλέπω, κυρία Λαγκάρτ. Έχω τρεις ε, δηλώσεις και να μου πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά που θα πω και αν όχι να μου εξηγήσετε γιατί. Είπατε μόνοι σας προηγουμένως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσει κανείς ε, τη διαφορά του 1,2% πληθωρισμού ή 1,8% παραδείγματος χάρη ενδεικτικά. Παρόλα αυτά, ε, παρά αυτό το επιχείρημα, το έολο θα έλεγα, ε, υπάρχουν ε, περίεργες πολιτικές ε, που εφαρμόζονται και συνεχίζονται. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Δεύτερον, βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον ε, στο βιομηχανοποιημένο κόσμο ε, τη μείωση της παραγωγικότητας ε, και παραμένουν πολλές φορές εταιρείε ζόμπι όπως αποκαλούνται. Τι είναι αυτές οι εταιρείε, Είναι εταιρείε που απλά επιβιώνουν λόγω των πολύ χαμηλών επιτοκίων. Με αυτές τις πολιτικές τελικά έχουμε μία αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες αναποτελεσματικές πλήρως και ως εκ τούτου όλες αυτές οι πολιτικές οδηγούν στην ε, χρηματοπιστωτική αστάθεια. Αυτές ήταν οι δηλώσεις μου. Ευχαριστώ. Μου δίνετε την ευκαιρία να διευκρινίσω αυτό που έλεγα και πριν για το 2%. Δεν είναι για να υποβάσω τη σημασία που έχει αυτή η συζήτηση. Οι παρατηρήσεις ε, είναι πολύ καλές, οδηγούν σε κάποιες προσδοκίες. Η συζήτηση μεταξύ εμπειρογνωμόνων, δηλαδή, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά ε, ο Κεντρικός Τραπεζίτης Αυστραλίας μιλούσε για μια ελάχιστη ευελιξία στην επίτευξη του στόχου για τον πληθωρισμό. Συνεχίζει τώρα στα αγγλικά, ενώ πριν μιλούσα γαλλικά η κυρία Λεγκάρ, δεν καταλαβαίνω γιατί μιλούσα γαλλικά και τώρα θα σας μιλήσω αγγλικά για τα υπόλοιπα. Από την άλλη λοιπόν αναφερθήκατε στο θέμα του πολύ χαμηλού κόστος χρηματοδότησης και αυτό διευκολύνει την επιβίωση εταιριών που αν δεν υπήρχε θα είχαν εξαφανιστεί. Ξέρετε και πάλι πρέπει να γίνεται ανάλυση κόστους ωφέλους. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτό το χαμηλό κόστος χρηματοδότησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ε, πόσα θα ήταν τα δάνεια, πόσες επιχειρήσεις θα χρηματοδοτούσαν τις δαπάνες τους. Υπάρχουν ε, πράγματα της ΕΚΤΟ όπως ο στοχευμένος μηχανισμός ε, χρηματοδότησης και αυτά έχουν στόχο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τώρα μπορούν να βελτιωθούν όλα αυτά τα εργαλεία έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος. Πιστεύω πως πράγματι μπορεί να υπάρξει μία εξειδίκευση. Και τώρα ξεκινάμε ε, στον τελευταίο γύρο των ερωτήσεων. Ε, τέσσερα λεπτά, ο Χωσέ Καρσία Μαργκάλ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, αγαπητή κυρία Λαγκάρτ. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω πάλι εδώ. Έρχεστε σε κάποια στιγμή διαφορετική από εκείνη που έφτασε ο κύριος Τράγκη το 2015 εν μέσω μιας υπαρξιακής κρίσης, με περιθώρια λιγμών όμως στην νομισματική πολιτική μέσω των επιτοκίων κλπ. Εσείς ε, φτάνετε όταν ο ήλιος μεν λάμπει, αλλά που υπάρχουν σύννεφα μαύρα στον ορίζοντα. Και όταν η νομισματική πολιτική έχει ήδη επιτόκια πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, ποια θα είναι η φύση της νέας κρίσης, θα είναι διαφορετική. Δεν θα είναι κρίση ζήτησης, αλλά κρίση προσφοράς από ό,τι φαίνεται. Οπότε ο ρόλος των διάφορων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας θα είναι διαφορετικός. Βραχυπρόθεσμα, όντω μπορούμε να παίξουμε με τη δημοσιονομική και την νομισματική πολιτική, αλλά πιο μακροπρόθεσμα χρειάζεται να έχουμε μεταρρυθμίσεις. Σας ρωτώ λοιπόν το εξή. Πόσο χρόνο πιστεύετε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία, για να μην μιλήσουμε για την παγκόσμια, μπορεί να συνεχίσει με αρνητικά επιτόκια χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα του συστήματος και τράπεζες. Δεύτερον, λαμβάνοντα υπόψη το ρόλο που θα παίξουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενεργητικού, ίσως θα έπρεπε να αλλάξουμε τον κανόνα που συνδέει την αγορά χρέους μιας χώρας ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας του και να αλλάξει και να υποφεληθούν οι χώρες οι οποίες χρωστούν. Έπειτα, η εμπειρία δείχνει ότι υπήρξε κάποια προτίμηση για τα ε, κρατικά ομόλογα. Μήπως θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερο πρωταγωνιστικό ρόλο στα, στο εταιρικό ενεργητικό. Μήπως θα ήταν λογικό το καλάθι των ενεργητικών που επιλέγονται να μεγαλώσει και να μην περιοριστούμε μόνο ε, στο τραπεζικό. Ευχαριστώ πολύ και Επαναλαμβάνω και πάλι, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, ελπίζοντας ότι θα αναλάβετε τα καθήκοντά σας επικεφαλής της ε, ΕΚΤ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σας δω και σε άλλες ε, συνθήκες. Λοιπόν, με ρωτάτε κάτι πολύ συγκεκριμένο, χωρίς να μπορώ εγώ να δώσω πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Πόσο καιρό θα έχουμε ακόμα αρνητικά επιτόκια. Μα δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Γιατί η σταθερότητα τιμών είναι το καθοριστικό. Τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν χρησιμοποιούνται πλήρως. Και ακόμα υπάρχει περιθώριο για να αναπτύξουμε κάποια από αυτά περισσότερο. Οπότε είναι δύνατο να πω τώρα πότε και κάτω από ποιες συνθήκες και πώς. Γιατί πρέπει να γίνει πρώτα μια ανάλυση κόστους-οφέλους ε, της χρήσης των μέσων αυτών. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μας και είναι νομίζω ότι το πρόγραμμα αγοράς θα παραμείνει ως έχει μέχρι να μην ε, ανέβουν τα επιτόκια. Ξέρω δηλαδή ποια σειρά θα ακολουθήσουμε. Οπότε αυτό βλέπουμε προς το παρόν. Τώρα, δεν ξέρω τι εννοείται μιλώντας για αγορά ομολόγων από τις εντός καλές ή λιγότερο καλές χώρες. Ε, δεν ξέρω αν εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε την ηθική μέσα σε αυτήν την άσκηση αντοχής. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τα κλειδιά της ΕΚΤ για να μπορεί να εκτιμήσει τι θα γίνει με τις αγορές αυτές. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει. Τέλο πάντων, μπορούμε να το συζητήσουμε ίσως αργότερα μεταξύ μας. Γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι αναφέρεστε στο σύστημα tiering, αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Ωραία. Εργίν Ερόγλου από το Renew, Παρακαλώ. Α, δεν είναι. Α, είναι εκεί, είναι. Αξιότιμη κυρία Λαγκάρτ, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Ε, τις τελευταίες δύο ώρες ε, τέθησαν αρκετά ερωτήματα, γι' αυτό ε, θέλω να εμβαθύνω κάτι, το θέμα των κρυπτονομισμάτων και των ψηφιακών νομισμάτων. Τα τελευταία χρόνια αυτά διαδίδονται όλο και περισσότερο και θέλω να ρωτήσω, αυτά αποτελούν ανταγωνισμό, ανταγωνιστικά νομίσματα στο ευρώ. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η και κατά πόσο είναι καθήκον της ΕΚΤ να αναχαιτήσει αυτή την εξέλιξη. Ε, ίσως ε, να δίδει και κάποιες συμβουλές ε, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και κάτι άλλο που δεν ετέθη σήμερα εδώ. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή η πολιτική της ΕΚΤ με τα αρνητικά επιτόκια αντιμετωπίζεται πολύ επικριτικά γιατί αυτή η πολιτική κυρίως ε, για τα μικρά ταμιευτήρια στη Γερμανία υπάρχει πρόβλημα. Κατά την άποψή σας ε, είναι απαραίτητο να υπάρξει συρρήκνωση του αριθμού των ε, τραπεζικών ιδρυμάτων ή θα μπορούσε στη Γερμανία να εκτιμήσει κανείς ότι με αυτή την πολιτική ενδεχομένως υπάρχουν ενδείξεις για μια επερχόμενη κρίση. Θα ήθελα ή δυνατόν να, μας, ε, να μου απαντήσετε. Φαντάζομαι δεν με ρωτάτε τι πιστεύω για μια συγκεκριμένη συγχώνευση τραπεζικών ιδρυμάτων. Λοιπόν, πάμε πίσω ε, στα ψηφιακά νομίσματα, ε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή καταρχήν ε, χρηματοπιστική σταθερότητα και αποφυγή και αποφυγή προβλημάτων. Ξέρετε, εγώ ε, θα ήθελα να διαφοροποιήσω τα διάφορα κρυπτονομίσματα που βεβαίως ε, αυτά αναλύονται διαφορετικά ανάλογα με το που ακριβώς ε, αντιμετωπίζονται. Υπάρχουν χώρες όπου αυτά τα νομίσματα αντιμετωπίζονται ως κεφάλαιο, ως ασφάλεια. Υπάρχει δηλαδή ένα ολόκληρο χάος για το σωστό πλαίσιο. Αλλά εντωμεταξύ έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ε, ιδιαίτερα μεταβλητό προϊόν, το οποίο όμως δεν απειλεί την σταθερότητα, δεν είναι εμπόδιο για την σωστή εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Εγώ αυτό θα το διαχώριζα από τα σταθερά νομίσματα, που κατά την άποψή μου είναι κάτι τελείως διαφορετικό και που ε, έχουν και διαφορετικό μέλλον. Βεβαίω, εγώ πιστεύω ότι τα σταθερά νομίσματα, είτε είναι λίμπρα είτε οτιδήποτε άλλο, η κεντρική τράπεζα ως προς τα ψηφιακά νομίσματα, αυτά τα ψηφιακά νομίσματα θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς. Δεν με απασχολεί τόσο κατά πόσον πρόκειται για τράπεζα ή όχι. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία η δραστηριότητα που αναπτύσσεται έτσι ώστε να διαφυλάσετε η συμμόρφωση με τους ε, κανόνες. Και γι' αυτό το λόγο εγώ θα έλεγα ότι οτιδήποτε μας προστατεύει από την ομοιοποίηση παράνομων εσόδων, από τη χρηματοδότηση της ε, τρομοκρατίας, από τη σωστή εφαρμογή των νομισματικών πολιτικών, όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οποτεδήποτε επιτραπεί να κυκλοφορούν αυτά τα νομίσματα εδώ αλλά και σε άλλες περιοχές. Γιατί χάρηκα όταν άκουσα ότι η ΕΚΤ εκλείπει από το G7 να εξετάσει τα ψηφιακά νομίσματα και να υποβάλει το στομό των δυνατών τα πορίσματά της. Ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Λαγκάρτ εγώ θέλω να σας πω, πριν από κάποιους μήνες ήμουνα παρόν στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ, μπροστά σε όλους τους ε, πολιτικούς ε, ομολόγησε ότι άκουσε υπερβολικά τις απόψεις ε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και έτσι εφαρμόστηκαν πολιτικές λιτότητες που μεταξύ άλλων γονάτισαν και τον ελληνικό λαό. Και σας ερωτώ, εφόσον ήταν σαφές ότι η κρίση του 2008 οφείλεται σε έλλειψη ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών, η οι οικονομολόγοι, οι θεωρητικοί, πολλοί από αυτούς αναφέρετε κι εσείς, εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι οι αγορές πρέπει να αυτορυθμίζονται. Και οι δυσλειτουργίες που υπάρχουν η ανισότητα για την οποία μιλήσατε προηγουμένως, αυτά οφείλονται ε, κυρίως ε, σε κακές πολιτικές και όχι στην έλλειψη των ρυθμίσεων. Εσείς μιλήσατε ότι δεν εφαρμόζονται οι συνθήκες και εγώ σας ερωτώ, ποια είναι η δική σας η άποψη ως προς το δεχόμενο το να αναθωρηθούν οι συνθήκες ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει μια νέα λειτουργία, δηλαδή να είναι το τελευταίο καταφύγιο για τις ε, διάφορες χώρες ανάλογα με τις ανάγκες τους και ως εκ τούτου στο καταστατικό ε, της ε, τράπεζας να είναι πρώτα απ' όλα η αντιμετώπιση της ανεργίας και όχι τόσο η σταθερότητα των τιμών. Well, any change to the... Οποιαδήποτε αλλαγή την εντολή της ΕΚΤ ε, εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εφεύρει η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν μπορούμε να περάσουμε από τη σταθερότητα των τιμών σε σταθερότητα των τιμών συν καταπολέμηση της ενεργείας, συν βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχει στο άρθρο 127 υποπαράγραφος 2 ένα σημείο το οποίο επιτρέπει στην ΕΚΤ ε, παράλληλα με την ε, ικανοποίηση του πρωταρχικού στόχου της σταθερότητας των τιμών να εξετάζει και τους δευτερογενείς στόχους που τίθενται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να διευκρινίσω και κάτι για μια προηγούμενη ερώτηση, ότι το περιβάλλον και η προστασία του περιβάλλοντος, αν θυμάμαι σωστά, είναι τμήμα αυτών των στόχων. Αυτό, επομένως, νομιμοποιεί την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ως δευτερογενούς στόχους που έχει πρωταρχική σημασία αλλά αποτελεί ένα δευτερογενή στόχο του, της ΕΚΤ. Δεν πρόκειται να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας για το ποιος έκανε τι σε σχέση με τα μνημόνια στην Ελλάδα. Πάντως και εδώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ιδίως στο τελευταίο τμήμα των προγραμμάτων, ε, έχει καταγραφεί ότι δήλωσε ότι οι απαιτήσει έναντι της Ελλάδος ήταν υπερβολικές σε σχέση σχέση με τις δυνατότητές και ότι το πρωτογενέ πλεόνασμα του 3,5% πρέπει να εγκαταληφθεί προ κάτι περισσότερο γραμμικό και πιο κοντά στο 1,5 έω 2% κατά μέγιστο. Ε, κοιτάξτε, υπήρχε η Τρόικα, λαμβάνονταν πολλές αποφάσεις από πολλούς φορείς. Δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο να αρχίσουμε να κατηγορούμε τον έναν ή τον άλλον. Ε, ήταν μια κοινή προσπάθεια. Και αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Η Ελλάδα μας είχε ζητήσει τη βοήθειά μας. Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή, αλλά είναι αλήθεια ότι υπέφερε λόγω του προγράμματος αναδιάρθρωσης που εφαρμόστηκε. Ευχαριστώ. Η την άλλη από τους Σοσιαλδημοκράτες. I can, but maybe not everybody. Το μικρόφωνο δεν είναι ανοιχτό. Okay. Thank you. So, a lot is... Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχει συζητηθεί πολύ το θέμα των πράσινων ομολόγων. Πολλά από τα προηγούμενα ερωτήματα αφορούσαν την πλευρά της συζήτηση. Όπως σωστά είπατε και στην απάντησή σας στις ερωτήσεις, ε, έχουμε πρόβλημα ε, προσφοράς. Και στο ερώτημα αυτό ανοίγεται και τη δυνατότητα δημόσιας παρέμβασης για να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο περιβάλλον για αυτή την αγορά. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Θα ήσασταν υπέρ ε, μιας μεγάλης δημόσιας έκδοσης πράσινων χρηματοπιστωτικών εργαλείων από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νομίζετε ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να υποστηρίξει αυτή την έκδοση, όχι αγοράζοντα την ιδιωτική αγορά που δεν ε, επιτρέπεται από τη συνθήκη, αλλά να τα δέχεται ε, ω εγγυήσει, δίνοντα προτεραιότητα σε αυτά τα ομόλογα σε σχέση με άλλου τύπου ομολόγων. Δεύτερο ερώτημα, τα κρυπτονομίσματα. Είπατε ότι δεν αποτελεί, αποτελούν απειλή ε, στα παραδοσιακά νομίσματα ή στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα το καλοκαίρι ακούστηκε η ιδέα ε, των κρυπτονομισμάτων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα αντίβαρο στην ηγεμονία του δολαρίου. Θα ήθελα να ακούσω το σχόλιο σας σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις και τι απαντήσεις θα μπορούσε να δώσει η ΕΚΤ σε αυτό. Ευχαριστώ. Για την πρώτη σας ερώτηση για τα πράσινα ομόλογα. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή, Επενδυτική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, είναι εκδότης τέτοιων ομολόγων και η ΕΚΤ στην ε, δευτερεύουσα αγορά αγοράζει κάποια τέτοια προϊόντα και το κατόφλι μέχρι το οποίο μπορεί ε, να έχει τέτοια ομόλογα δεν είναι 33% αλλά 50% ναι. άρα τις επιτρέπεται να έχει ε, περισσότερα βράσινα ε, ομόλογα σε σχέση με άλλα ομόλογα και αυτό είναι θετικό. Επίσης χαίρομαι διότι η Ursula von der Leyen προωθεί ενεργά μία νέα πράσινη συμφωνία. Είναι της γνώμης ότι η έκδοση αυτών των ομολόγων έχει κέρια σημασία και συμφωνώ απολύτως. Για τα κρυπτονομίσματα και για την πρόταση του Μακάνη. Με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ. Μου κίνησε το ενδιαφέρον η πρόταση αυτή. Δεδομένων των συνεχών εξελίξεων. Με δύο λόγια να πω για αυτούς που δεν διάβασαν την ομιλία του Μακάνη, αυτό που προτείνει είναι κάποιες από τις βασικές κεντρικές τράπεζες να σχηματίσουν ε, μια κοινοπραξία και να διερευνήσουν κατά πόσο είναι δυνατόν να δημιουργήσουν ε, νομίσματα των κεντρικών τραπεζών, κοινά νομίσματα. Αυτό που έχει κατά νου ε, το Λίμπρα δηλαδή, αυτοί που επινόησαν το Λίμπρα, να υπάρχει ένα εργαλείο μετατρέψιμο ε, σε κρατικά νομίσματα. Ο Μακάνη προτείνει κάτι παρόμοιο, αλλά θα είναι κάτι το, θα το οποίο θα εκδίδουν οι ίδιες οι κεντρικές τράπεζες. Και όντως ε, αυτό έχει αρκετές ενδιαφέρουσες πτυχές. Μπορούμε να τις διερευνήσουμε. Δεν μπορώ να προδικάσω ποια θα είναι η άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, αλλά προσωπικά θα ήθελα να συμμετάσχω σε μια τέτοια διερεύνηση αυτής της νέας έννοιας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ εκπροσωπώ τους πολίτες μιας χώρας που δεν είναι στην Ευρωζώνη, την Ουγγαρία και θέλω να σε ρωτήσω το Πρώτον, για τη συνεργασία μεταξύ χωρών Ευρωζώνη, χώρε χωρίς τη Ευρωζώνη. Είναι ζωτική σημασία να υπάρχει μια καλή συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών χωρών. Ό,τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη επηρεάζει πάρα πολύ τις χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Ε, είναι αυτό που λέμε ότι βύχης ε, στην Ευρωζώνη παθαίνει πνευμονία ε, κάποιος που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Οπότε θέλω να το ξέρετε αυτό. Υπάρχει μια νέα πρόταση η οποία εγκρίθηκε εν μέρη για την δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης και σίγουρα το γνωρίζετε ότι έχουν δημιουργηθεί πολλές ανησυχίες στις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Στη γραπτή σας απάντηση είπατε ότι σα σας ικανοποιεί μια τέτοια πρόταση. Οπότε πώς σχεδιάζετε να αντιμετωπίσετε τις ανησυχίες αυτές που εκφράζουν οι χώρες που δεν είναι στο ευρώ, που δεν έχουν το ευρώ. Και τι γίνεται με τις προποθέσει ένταξη στην Ευρωζώνη. Γιατί υπάρχουν ότι προηγουμένως πρέπει να συμμετέχουν σε δομές κτλ. Οπότε θέλω να ρωτήσω, οι προποθέσει που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα είναι επαρκής ή νομίζετε ότι θα δημιουργήσετε και άλλες προϋποθέσεις. Γιατί έτσι θα ξέρουμε και εμείς αν απεξερχόμαστε επαρκώς στις υποχρεώσεις μας και είμαστε έτοιμοι ή όχι να μπούμε. Τέλος, για τα μαθήματα που έχουμε πάρει από την τελευταία κρίση, η χώρα μας χρησιμοποίησε η Ουγγαρία ε, μεικτά μέσα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση ε, πολλά από αυτά βέβαια δεν άρεσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φαίνεται ότι λειτουργήσαν. Γιατί για δεύτερη χρονιά η Ουγγαρία έχει την μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Ήδη εσείς είπατε ότι ήταν πολύ καλή δράση της ΕΚΤΑ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, τι πιστεύετε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά και οι χώρες μέλη για να αποφύγουν μια νέα απειλή, μια νέα κρίση. Τι θα πρέπει να γίνει διαφορετικά τώρα από τις χώρες μέλη για να αποφευχθεί μια πολύ χαμηλότερη ανάκαμψη στην Ευρωζώνη σε σχέση με αλλού. Απάντηση. Η συνεργασία ανάμεσα στις χώρες Ευρωζώνης και μη Ευρωζώνης είναι πάρα πολύ σημαντική, το πιστεύω και εγώ αυτό. η επιθυμία είναι να είναι 26 εκτός από τις χώρες opt-out, Δανία και ελπίζουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να λύσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο το θέμα του. Η συνεργασία λοιπόν είναι ζωτική σημασία γιατί είμαστε όλοι μέλη τη ίδια οικογένεια. Θα ζούμε μαζί. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική πράγματι. Ναι, όντω. Καλωσόρισα την εμβρυγική μορφή της δημοσιονομικής ικανότητας που αναφέρθηκε τον Ιούλιο ε, και την ε, καλωσορίζω, τη βλέπω θετικά σαν ένα πρώτο βήμα, γιατί μπορεί να βοηθήσει στη σύγκληση κλπ. Αλλά ίσως να πρέπει να πάμε ακόμα πιο μακριά, εφόσον οι προϋποθέσεις το επιτρέπουν και οι χώρες μπορούν να ακολουθήσουν. Και πάλι λοιπόν η συνεργασία με τις χώρες εκτός Ευρωζώνης είναι σημαντική, γιατί κάποια στιγμή θα μπουν σε αυτή την ομάδα. Ελπίζω να προχωρήσουμε κάτω από τις σωστές προϋποθέσεις. Επιπλέον προϋποθέσεις ε, για να μπορούν να ενταχθούν ε, οι χώρες στο ευρώ. Το είδαμε και στην περίπτωση της Κροατίας ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Μπαίνουν στην ε, Τραπεζική Ένωση, τηρούν τις αρχές, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Εγώ προσωπικά Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει πρόοδος στο θέμα της καταπολέμησης νομιμοποίησης ε, χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες και αντιμετώπιση και καταπολέμηση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών. Δεν λέω ότι αυτά που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας αρκούν. Πρέπει να γίνουν περισσότερα και σίγουρα βοηθάει η συνεργασία. Ο κ. Παπαδημούλης, παρακαλώ. Ε, σας καλωσορίζω κυρία Λαγκάρτ. Σημειώνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση όσα είπατε για την ανάγκη να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια για τη χώρα μου. Και σημειώνω επίσης με ικανοποίηση την επισήμανσή σας ότι η ελληνική οικονομία σημειώνει μια ισχυρή ανάκαμψη το τελευταίο διάστημα, πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Πριν λίγο δόθηκαν τα επίσημα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2019 με μια ανάπτυξη 1,9%. Ελπίζω την πρότασή σας να την ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργό, ο νέος Έλληνας Πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης, έτσι ώστε να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η χώρα μου, ε, συζητώντας με τους δανειστές, για πιο χαμηλά ρεαλιστικά πλεονάσματα. Ελπίζω να είναι το ίδιο φιλόδοξος με εσά σε αυτή τη διεκδίκηση. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, όμως και για όσα υπέφερε η χώρα μου και ο λαός μου, ιδιαίτερα στα πρώτα δύο μνημόνια. Ο κύριος Ντομινίκ Στροσκάν, ο κύριος Ντάισεμπλουμ, μίλησαν για τους περίφημους λάθος πολλαπλασιαστές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που προκάλεσαν τριπλάσια ανεργία, και μια ύφεση διπλάσια αυτών που υπολογίζατε ως Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είπαν με θάρρος ότι αυτά έγιναν, όπως και η μία αναδιάρθρωση του χρέους, για να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των γαλλικών και γερμανικών τραπεζών. Εσείς ποια γνώμη έχετε, γιατί οι δύο κύριοι που ανέφερα είναι τέος πλέον. Εσείς εφαρμόζετε ένα παράδειγμα ανακύκλωσης. Περνάτε από την ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα είχε λοιπόν σημασία να μας πείτε τη γνώμη σας, γιατί το κουτί της Πανδώρας άνοιξε πριν από πολλά χρόνια σε βάρος της χώρας μου και δεν θα ανοίξει τώρα αν είμαστε όλοι ειλικρινείς. Και το δεύτερο που θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω, επειδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να έχει περισσότερη διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία από το Ευρω... Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για να ενισχύσετε αυτή τη διαφάνεια. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παπαδημούλη. Νομίζω ότι αυτά που είχα να πω για το πρωτογενές πλεόνασμα στην Ελλάδα τα είπα. Και είπα επίσης ε, το πόσο αγωνιστήκαμε για να περάσουμε τη δική μας τη θέση. Τη δική μου τη θέση που ήταν διαφορετική. Ε, γι' αυτό το λόγο ε, δεν θελήσαμε να αλλάξουμε στην τρίτη φάση του προγράμματος. Πράγματι, είναι αλήθεια, πολλές από τις ε, διαρθρωτικές αλλαγές ήταν ένα κομμάτι του συνολικού πακέτου και εκεί ε, δεν υπήρξε ε, σωστή εφαρμογή. Θέλω να ελπίζω ότι η νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα θα συνεχίσει αυτά που έχουν ήδη ξεκινήσει, θα εμβαθύνει όμως περισσότερο, ε, θα καταστήσει την ε, Ελλάδα ανταγωνιστικότερη. Εγώ χαίρομαι που υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα και χαίρομαι ε, που στην Ελλάδα πλέον ξεκινάνε περισσότερες τουριστικές αλλά και μεταποιητικές δραστηριότητες. Όσον αφορά τον δημοσιονομικό συντελεστή, τον πολλαπλασιαστή μάλλον, το αναγνωρίσαμε αυτό, όχι μόνο σε σχέση με εσά, αλλά και σε σχέση με την Πορτογαλία. Τότε που εξετάσαμε τι επιπτώσει του πολλαπλασιαστή στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Αναγνωρίσαμε ότι είχαμε υποεκτιμήσει, υποτιμήσει ε, τι επιπτώσεις από τον πολλαπλασιαστή και γι' αυτό θελήσαμε να προσαρμόσουμε τα μέτρα ε, που θα έπρεπε να ληφθούν ε, βάσει του προγράμματο. Πράγματι, δεν ήταν όμως ευθύνη ενός μόνο ή δύο οργανισμών, όλοι έφεραν κατά κάποιον τρόπο την ευθύνη και γι' αυτό δεν έχει νόημα τώρα να αποδίδει κανείς ε, υπετιότητες. Είναι βέβαια σημαντικό να αναγνωρίζει κανείς όταν κάτι δεν είναι σωστά σχεδιασμένο ε, να το αναγνωρίζει και νομίζω ότι εμείς ε, το κάναμε με απόλυτη σαφήνεια. Εμείς έχουμε ένα εσωτερικό μηχανισμό, έχουμε ένα γραφείο που κάνει εσωτερικές αξιολογήσεις και εκεί λοιπόν έχει συζητηθεί επανειλημμένα το θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα στη διαφάνεια, εγώ είμαι στο να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια που να είναι και συμβατή με την ανεξαρτησία του θεσμού. Ε, όμως θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι η συζήτηση που θα γίνει, αν τελικά ε, οριστό, διοριστό, ε, τέσσερις φορές το χρόνο, πέντε φορές με την Επιτροπή και μία φορά στην Ολομέλεια, όλα αυτά θα είναι ένα κομμάτι της διαφάνειας υπέρ της οποίας ε, τάσσομαι ανεπιφύλακτα. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε άλλες πέντε ερωτήσεις και άλλε δύο ερωτήσει στο κάτσι. Αν δεν τελειώσουμε στη μία, θα συνεχίσουμε μετά τη μία στα αγγλικά για να μπορέσετε κι εσεί, ε, κύριε Λαγκάρτ, να ε, κάνετε την καταληκτική σα παρέμβαση. Ίσως μπορούμε να τελειώσουμε μία και πέντε, αν είσαστε αρκετά γρήγοροι ε, και αν είσαστε και πιο στοχευμένοι. Ιωαχήμ Σούστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν τεθεί πάρα πολλέ ερωτήσει, γι' αυτό και εγώ θα περιστώ σε δύο μόνο θέματα. Αφενό, ε, για μένα είναι αυτονόητο ότι πρέπει να συνεχίσουμε την πολιτική των χαμηλών επιτοκίων τη στιγμή που πάρα πολλά κράτη εφαρμόζουν μια περιοριστική ε, δημοσιονομική πολιτική. Βέβαια, αυτή η πολιτική τη Κεντρική Τράπεζα έχει και αρνητικέ επιπτώσει, παραδείγματο χάνει στα αρνητικά επιτόκια. Τώρα στη Γερμανία ε, έγινε μια πρόταση από ένα συγκεκριμένο κόμμα όπου λένε ε, από τον νόμο να απαγορεύεται οι τράπεζες ε, να εξακολουθούν να εφαρμόζουν αρνητικά επιτόκια σε καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Εσείς αυτό το βρίσκετε σωστό ή τι έχετε να μας πείτε. Κατόπιν, όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων στην ε, Ευρωζώνη, το αποτέλεσμα των συζητήσεων είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά επιτόκια σε διάφορα κράτη. Αυτό όμω είναι ανόητο, διότι έχουμε κράτη με υψηλότερο δανεισμό και με τον τρόπο αυτό έχουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα οι χώρε αυτέ να αποπληρώσουν τα χρέη του. Και μόνο αυτό, αλλά αποδυναμώνεται και το ευρώ. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ στο πλαίσιο του να υπάρχει ένα ενιαίο νομισματικό χώρο και μια ενιαία κοινή αγορά. Ε, δεν είναι αυταπάτη το να θέλει κανείς να αποφύγει την κοινή διαχείριση κινδύνων. Και μία ερώτηση, τι μέτρα θέλετε να λάβετε έτσι ώστε στην Ευρωζώνη υπάρχει πραγματικά μία δίκαιη διαχείριση κινδύνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συνδέετε τα επιτόκια και την δημοσιονομική πολιτική που πρέπει να εφαρμόσουν κάποια κράτη-μέλη. Νομίζω ότι όλα εντάσσονται στην ίδια συζήτηση και όλα αυτά εκφράζουν και αυτά που ε, λένε κεντρικοί τραπεζίτες, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, διάλογος έτσι ώστε ε, να μπορεί να μετρηθεί το κόστος και το όφελος μέτρων τα οποία είναι απαραίτητα έτσι ώστε να φτάσει κανείς και στην επιθυμούμενη σταθερότητα τιμών. Επίσης πιστεύω ότι κάποια μακροπροληπτικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται για να αντιμετωπίζονται κίνδυνοι είναι σε συγκεκριμένους τομείς. Αυτά πρέπει να συνεχίσουν ε, και πρέπει ε, να ε, εφαρμόζονται όταν υπάρχει αστάθεια. Πρέπει να σας πω, ανησυχώ ιδιαίτερα σχετικά με το θέμα της μόχλευσης των δανείων. Προφανώς ε, πολλοί τραπεζίτες εστιάζουν σε αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να το ελέγχουμε πολύ προσεκτικά για να μπορέσουμε να αποφύγουμε την ε, διαμόρφωση κινδύνων. Ε, υπάρχουν τα κάποια μακροπροληπτικά εργαλεία, αλλά θα πρέπει και αυτά να ε, χρησιμοποιούνται σωστά. Καλύτερη διαχείριση κινδύνων στην ε, Ευρωζώνη, αυτός είναι ο τελικός στόχος, διότι η Νομισματική Ένωση θα πρέπει να αφορά ε, τόσο τους κινδύνους, όσο και την κοινή διαχείριση της ε, επιβράβευσης αν θέλετε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα βέβαια σε αυτό το σημείο. Η Ευρωζώνη ακόμα δεν έχει εκπληρώσει όλους τους, τους στόχους. Υπάρχουν ακόμα κάποια που υπολείπονται. Αν δείτε λιγάκι το θέμα των απολόγων σε διάφορες, κάθε μία χώρα, βλέπουμε ότι ε, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στην απόδοση και είναι εντυπωσιακό το πώς ε, τα τελευταία τρίμηνα υπήρξε και μία σύσφυξη. Τώρα, είναι αυτός ο δρόμος προς ε, ένα ελάχιστο spread που είναι αποδεκτό για να υπάρχει διαχείριση και εξάπλωση κινδύνων. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση και όπως ανέφερε σήμερα το πρωί ο κύριος Ενρία να ολοκληρωθεί το θέμα των κόκκινων δανείων, αυτά που συνεπάγονται στους ισολογισμούς. Πρέπει να γίνει ακόμα πολλή δουλειά πριν ακόμα περάσουμε στην κοινή διαχείριση κινδύνων, κάτι στο οποίο αναφερθήκατε και που θα ήταν ιδανικό αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Πρέπει όμως να δουλέψουμε πάνω στις προϋποθέσεις για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να μετακινηθούμε στη σωστή κατεύθυνση. Κύριο thank uh, ούτε από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαγκάρντ. Ίσως αποφύγαμε τα χειρότερα, δηλαδή να μπουν επικεφαλής της ΕΚΤ ε, ε, αυτούς που είναι λαϊκιστές. Με το οικονομικό σενάριο ε, που έχουμε τώρα, θα χρησιμοποιηθεί η εργαλειοθήκη που μέχρι τώρα χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στο παρελθόν. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά τις παρενέργειες αυτών των πολιτικών που πρέπει να εξεταστούν. Σε προηγούμενη απάντησή σας ε, αναφέρατε ε, τις ε, επιπτώσεις στην αγορά κινήτων. Έχουν αυξηθεί οι τιμές των ακινήτων και είναι πραγματικό πρόβλημα για τις πόλεις μας η πολιτική της μη αύξησης των επιτοκίων είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά θα πρέπει και να αντισταθμίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις. Τι να κάνουμε με τα μακροπροληπτικά ρυθμιστικά εργαλεία, όπως είπατε πριν. Είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τα αντικυκλικά προστατευτικά μέτρα και άλλες εγγύησεις για να αντισταθμίσετε τα αρνητικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Για το συγκεκριμένο αυτό τομέα, τα ε, μακροπροληπτικά εργαλεία τα οποία πρόσφατα χρησιμοποιήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν δείξει την αποτελεσματικότητά τους για την αγορά κινήτων. Αν δείτε πώς επηρεάστηκε η αγορά κινήτων στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε διάφορες χώρες όπως αυτές, όπου υπήρχε μια έκρηξη των τιμών στην αγορά κινήτων, τα εργαλεία μακροπροληπτικά, είτε είναι δείκτης δανείων προς εισόδημα, είτε κάτι άλλο, ήταν αποτελεσματικά και πρέπει να χρησιμοποιούνται. Στις παρούσες συνθήκες νομίζω ότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται. Και να προσθέσω πολύ σύντομα ότι πιστεύω ότι είναι και θέμα προσφοράς. θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών και ίσως να μπορεί να διευκολυνθεί αυτός ο τομέας, ίσως και με δημόσιες επενδύσεις. Αντώνιο Ρινάλδη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαγκάρντ. διεξάγεται μια συζήτηση σε σχέση με την έντολη της ΕΚΤ και σε σχέση με τις δημοσιοποιήσεις στοιχείων. Και απαντήσατε και σε προηγούμενη ερώτηση συναδέλφου. Είπατε ότι ο πρωτογενής στόχος της ΕΚΤ είναι η σταθερότητα των τιμών και η αποφυγή του πληθωρισμού. Αλλά και πολλοί εθνικοί φορείς θεωρούν την απασχόληση ως πρωταρχικό στόχο. ίσως ο στόχος της ε, απασχόλησης να μπορέσει να αποτελέσει πρωταρχικό στόχο. Αυτή την ερώτηση θέλω να σας θέσω, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτή τη χρονική στιγμή. Ένα δεύτερο ερώτημα. Μπορείτε αυτή τη χρονική στιγμή να εγγυηθείτε στους πολίτες της Ευρώπης την απόλυτη ανεξαρτησία σας. Και αυτό το ερωτώ ως απλός πολίτης της Ευρώπης. Τον Ιούνιο του 2013, όταν δημοσιεύτηκε αυτή η επιστολή στη Λεμόντ, είπατε ότι δεν θέλουμε καν να τα ακούσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αν εγώ γίνω ε, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε, ε, τότε είπατε στον κύριο Σαρκοζή, χωρίς ε, την ε, κατεύθυνση θα είμαστε αναποτελεσματικοί, δεν θα είμαστε αξιόπιστοι. Έχουμε ανάγκη έναν άνθρωπο στην αρχή της ΕΚΤ που να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστος και ανεξάρτητος. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ να μας διαβεβαιώσετε ότι εσείς σε αυτή τη θέση θα είσαστε απόλυτα ανεξάρτητοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Γιατί νομίζω για το θέμα της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας ε, και για το θέμα της ανεξαρτησίας ε, του Προέδρου της ΕΚΤ, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι ναι, πιστεύω ότι συνδέεται εν με την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της Κεντρικής Τράπεζας. Σε πολιτικά περιβάλλοντα, αν ανήκει κανείς στο γραφείο ενός υπουργού, αν ε, λειτουργεί μόνος του και δεν έχει την υποστήριξη του ηγέτη, δεν έχει επαρκή αξιοπιστία. Στην περίπτωση του Προέδρου της ΕΚΤ, αυτό το βλέπω ως εντελώς διαφορετική, διαφορετική περίσταση και είναι κάτι ε, το οποίο το παρέχει και ο νόμος. Ε, ο νόμος ζητάει από τους ηγέτες των κρατών μελών να μην ασκούν πίεση στον επικεφαλής της ΕΚΤ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένα θεσμικό όργανο που υπηρετεί τους πολίτες της Ευρωζώνης και όχι τους ηγέτες των κρατών μελών και λογοδετεί στους πολίτες της Ευρωζώνης μέσω ημών που είστε οι εκπρόσωποι των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, κατ' εμέ λοιπόν είναι κέρια σημασία αυτό και χωρίς αυτή την ανεξαρτησία δεν θα είχα καν σκεφτεί να υποβάλω υποψηφιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Στη διαδικασία του Catch the Eye, δύο ερωτήσεις. Θα μιλήσω γαλλικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ε, παρέμβασή σας. Χαίρομαι για την υποψηφιότητά σας για την Προεδρία της ΕΚΤ η αξιοπιστία που ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι και γιατί είστε και η πρώτη γυναίκα υποψήφια. Σήμερα είμαστε πέντε γυναίκες από τους 24 ομιλητές που έλαβαν το λόγο. Καμιά φορά η ποιότητα υπερισχύει της ποσότητας. Ούκεν το πολλό το εφ. Εγώ είμαι από την Νορμανδία νομίζω όπως και εσείς κυρία Λαγκάρντ. Και νομίζω ότι οι μεγάλες ε, ε, αλλαγές για το κλίμα, για την τεχνολογία και για άλλα θέματα, μας υποχρεώνουν να επανεξετάσουμε την οικονομική και νομισματοπιστωτική στρατηγική μας. Το ερωτηματολόγιο ε, με τις απαντήσεις σας δείχνετε ότι ε, σκέφτεστε ε, την επανεξέταση της θέσης της ΕΚΤ έναντι των πολιτών, ώστε να ακούτε περισσότερο τη γνώμη των νέων και της κοινωνίας των πολιτών στην ε, Επιτροπή μας ε, θέλουμε μια νομισματική πολιτική που να ε, υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα συμφέροντα των καταναλωτών, γιατί οι καταναλωτές είναι οι βασικοί οικονομικοί παράγοντες. Για όλα αυτά λοιπόν, πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε τη δράση της ΕΚΤ περισσότερο κατανοητή, περισσότερο συγκεκριμένη και περισσότερο ανοιχτή παραδείγματο χάρη μέσω των ετησίων φόρουμ που πρότεινε κάποιο συνάδελφο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Χαιρετίζω την Αντιπρόεδρο και ως γυναίκα και ως ε, καταγόμενη από την Ορμανδία, όπως είπατε. Τα ετήσια φόρουμ που αναφέρθηκαν είναι όντως ένας τρόπος να συμπεριλάβουμε την κοινωνία των πολιτών, αλλά νομίζω ότι δεν αρκεί αυτό. Και πιστεύω συγκεκριμένα ότι για να μπορέσουν τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωζώνης ε, να πάρουν στα χέρια τους αυτή την πολιτική, πρέπει να περάσουμε από όλα τα κανάλια που φτάνουν προς αυτούς, με όλες τις γλώσσες που είναι κατανοητές ε, προς αυτούς στο Διεθνές Ομισματικό Ταμείο ζήτησα από όλους τους συνεργάτες μου να σταματήσουν να χρησιμοποιούν συντομογραφίες γιατί ε, χρησιμοποιώντας τα αρχικά οργανισμών απομονώνουν τους πολίτες που δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα που μιλάμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε μέσω της γλώσσας μας να απευθυνθούμε προς πολίτες, προς καταναλωτές που δεν είναι εμπειρογνώμονες ε, σε θέματα νομισματικής πολιτικής, να καταλάβουν τι είναι η έκτηση, τι χρησιμεύει, ε, γιατί ε, αποτελεί ένα στοιχείο περιφερειακής κυριαρχίας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όλα αυτά είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν και πιστεύω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα θελήσει με τα χαράς να προχωρήσει σε μια διαφορετική προσέγγιση και πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να γίνει. Okay, now the last speaker, last... Τελευταία ερώτηση. Κούσμαν. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Εδώ είμαι δεν είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει δύναμη. Καλά να μιλήσω αγγλικά τότε. Should respect limit for, for interpreters. Uh, I agree with uh, many of my... Συμφωνώ με πολλούς από τους συναδέρφους που είπαν ότι η μη συμβατική νομισματική πολιτική ήταν αναγκαία για να αποφευθεί η κατάρρευση της Ευρωζώνης. Και συμφωνώ επίσης ότι η μη συμβατική νομισματική πολιτική ελοχεύει και κινδύνους. Θέλω λοιπόν να βασιστώ στην εμπειρία της δικιάς μου χώρας που είχαμε ένα πακέτο λιτότητας ε, με νομισματική παρέμβαση στην Πορτογαλία που οδήγησε σε πολύ μεγάλη ύφεση αλλά επιπλέον και σε μεγάλη αύξηση του χρέους αυτά τα χρόνια της λιτότητας. Τα προηγούμενα χρόνια η νέα πολιτική πλειοψηφία αντέστρεψε τα μέτρα και έτσι είχαμε τα καλύτερα χρόνια σε ανάπτυξη όσον αφορά τα χρόνια που είμαστε εμείς στο ευρώ, αλλά και την μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους. Οπότε, η συζήτηση που πρέπει να γίνει, και αυτή είναι και η ερώτηση που σας μεταφέρω, είναι το εξή. Πιστεύετε ότι αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους της ε, ε, πολιτικής ε, μη συμβατικών μέτρων μήπως ε, οδηγεί σε ένα νέο προβληματισμό ή πιστεύετε ότι η σταθερότητα της Ευρωζώνης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με νομισματική πολιτική που συνδυάζεται με πολιτικές λιτότητας όπως είχαμε μέχρι τώρα. Μπορεί είναι καλύτερα δηλαδή να έχουμε κάποιο μείγμα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να χαιρετήσω τις προσπάθειες της Πορτογαλίας και των γάλλον που πέρασαν από μια τόσο δύσκολη περίοδο. Και δεν με εκπλήσει το ότι ε, η αναλογία ΑΕΠ χρέους βελτιώθηκε πάρα πολύ, γιατί άρχισε να αναπτύσσεται η Πορτογαλία βγαίνοντας από το πρόγραμμα. Και οι συνάδελφοι στο Δούνου του λένε ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία, παρόλο που βέβαια για τρία χρόνια ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και χρειάστηκε να γίνουν πολλές μεταρρυθμίσει. Πάντως και συμβαίνει συχνά όταν έχουμε πολιτικές αλλαγέ, Οι επόμενοι ακολουθούν μετά από το σημείο δηλαδή που σταμάτησαν οι προηγούμενοι. Και εκείνοι υποφελούνται από τα θετικά αποτελέσματα. Πάντως ήταν πολύ θετικέ οι εξελίξει. Πάντως, διαφωνώ μαζί σας για το ότι οτιδήποτε εξωτερική τριγμή για την Ευρωζώνη ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να χρησιμοποιεί το μείγμα που λέτε. Σίγουρα χρειάζονται και μεταρρυθμίσεις που είτε ήδη γίνονται ή πρέπει να γίνουν περισσότερες. Πιστεύω δηλαδή τελικά ότι αυτά πρέπει να βγαίνουν μαζί και με αυτό θα τελειώσω και δεν θέλω να σας επιβάλλω επιπλέον δύο λεπτά. Η συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της Ευρωζώνης, βάζοντας στο κέντρο τον άνθρωπο, είναι ε, αυτό που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και αυτό θα κάνω και εγώ ως επικεφαλής της ΕΚΤ. Είμαι έτοιμη να το κάνω